Ladies, gentlemen, colleagues, we need to get started. We... να Ήδη έχουμε μου να αρχίσω με την ακρόαση την οποία που έχουμε, την εμπορική συμφωνία Ευρωξένους Κολομβίας και Περού. Με τη συμμετοχή του Επιτρόπου Αρμοδίου για το Εμπόριο, Καρέλ Ντεγκούχτ. Όπως ξέρετε, άρχισε αυτή η συμφωνία το Μάρτιο πέρσι. Και σήμερα βρίσκεται στο Συμβούλιο, η τελική υπογραφή προβλέπεται τον Απρίλιο, μετά από τις αποφάσεις θα λάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνέντευξη εδώ σύμφωνα με την συνθήκη της Λισαβόνας για τη σύναψη συμφωνίας με τρίτες χώρες. Αυτή η διαδικασία προβλέπει να ολοκληρωθεί φέτος το φθινόπωρο. Η ακρόαση αυτή αρχίζει μία διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ε, καλωσορίσω όλους τους ομιλητές και κυρίως αντιπροέδρους του Περού και της Κολομβίας που είναι παρόντος. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους εμπειρογνώμονες. Πρώτα απ' όλα, θα ακούσουμε τον κύριο Αντριάν Βαντενχόβεν, διευθυντή των ε, τμήματος διεθνών ε, σχέσεων του Business Europe, που εκπροσωπεί τις ε, ενώσεις επιχειρηματιών της Ευρώπης. Αντριάν, σε καλωσορίζουμε. Τον Ερντοάδο Εστέβεθ, σύμβουλο της Τούκα, τον Οράσιο Κουιντό, που είναι συντονιστής της Διεθνούς Ένωσης για τις λογικέ Συμβάσεις από το ΕΛΟ και τελικά τον Επίτροπο Καρέλ Ντεγκούχ, τον οποίο καλωσορίζω. Και βεβαίως θα ήθελα να καλωσορίσω τον Αντιπρόεδρο της Κολομβίας, Αγχελίνο Γκαρθών, και την Αντιπρόεδρο Μαρισόλε Σπινόσα από το Περού που βρίσκεται στο Προεδρείο αριστερά μου. Σύμφωνα με τους εξής κανόνες θα γίνει αυτή η ακρόαση. Δεδομένου ότι έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, προτείνω όλες οι παρεμβάσεις από τους συμμετέχοντες να περιοριστούν σε 2-3 λεπτά. Και το εννοώ 2 με 3 λεπτά. Διότι είμαστε εδώ για να ακούσουμε τους εμπειρογνώμενες και όχι τους συναδέλφους. Σας παρακαλώ λοιπόν, εάν θέλετε να λάβετε το λόγο, να το πείτε στη γραμματεία για να κανονίσουμε τον χρόνο ομιλίας. Αρχίζουμε λοιπόν με τους συμμετέχοντες. Έχουν 7 λεπτά. minutes, I'll indicate that they have minute left. This applies to... Όταν πλησιάζει ο χρόνος που έχουν στη θέση του στο τέλος, ένα λεπτό πριν, να χτυπήσω το καμπανάκι για να το ξέρουν. Θα ολοκληρώσω τον πρώτο κύκλο. Ο Επίτροπος για 10 λεπτά και αρχίζουμε. Με τον Αντριάν Χόβεν. Ορίστε, παρακαλώ. Thank you, Mr. Chairman. Thank Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητά μέλη αυτής της Επιτροπής. Είναι τιμή μου χαρά μου για μένα που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να εκφράσω την υποστήριξή μας ε, ως προς την έγκριση αυτών των ε, συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου. Είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση το να συνεχίσει τη συνεργασία της με την Κολομβία και το Περού και μάλιστα με έναν ισόρροπο τρόπο έτσι ώστε να λαμβάνει η συμφωνία υπόψη της ε, τις δυνατότητες που υπάρχουν και με ρεαλιστικό τρόπο να λαμβάνει υπόψη της τις επιταγές της περιφερειακής οικονομικές αλλά και τι πολιτικέ αυτών των χωρών. Επιτρέψτε μου καταρχήν να επισημάνω γιατί είναι σημαντικό για τι ε, ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. να ε, εμπλακούν στη διαπραγματεύση ελεύθερου εμπορίου με τις χώρες αυτές. Πρώτον, όλοι γνωρίζουν ότι στις αγορές αυτές υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός από τις ΗΠΑ από την Ασία, από παίκτες της Ασίας στην παγκόσμια αγορά. Κατόπιν τούτου, αυτή η μορφή συμφωνία προσφέρει στις ευρωπαϊκέ επιχειρήσει τη δυνατότητα να αναπτύξουν περισσότερε σχέσει στην περιοχή. Αυτό είναι σημαντικό, διότι σήμερα βλέπουμε ότι στην Κολομβία και στο Περού έχουμε υψηλό βαθμό ανάπτυξης και ε, ε, προβλέπονται πολλές επενδύσεις σε σημαντικούς κλάδους ε, όπου είναι ισχυρή η ευρωπαϊκή βιομηχανία όπως τον τομέα της ενέργειας. Νομίζω πολλές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την τεχνολογία στην Ευρώπη θα επενδύσουν και αυτές. Επίσης προβλέπονται επενδύσεις στον τομέα της υποδομής αλλά θεωρώ και πάλι ότι θα ήταν καλό οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε ορισμένα από αυτά τα προγράμματα. Το θέμα όμω δεν είναι μόνο οι επενδύσεις, είναι και το παραδοσιακό εμπόριο. Και στο σημείο αυτό μπορούμε να ευχαριστήσουμε τους διαπραγματευτές ε, για αυτά που έχουν κάνει για το βιομηχανικό στοιχείο των διαπραγματεύσεων που αποδείχθηκε ιδιαίτερα επωφελές για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Υπάρχουν ορισμένα θέματα, θα τα προβάλλω σημαντικά από βιομηχανική πλευρά. Το ένα είναι οι κανονισμοί κυρίως στην Κολομβία για τα βιοκαύσιμα και η αναγκαιότητα να υπάρξουν διαβουλεύσεις με Ευρωπαίους παραγωγούς άνθρακα για το ποιες προδιαγραφές θα ισχύουν. Γιατί οι αυτοκινητοβιομηχανίες πρέπει να γνωρίζουν τα συστήματα εσωτερικής κάψης ε, για να προσαρμοστούν. Κάτι άλλο αφορά την ε, ένδυση και την κλωστεφαντουργία. Είναι σημαντικό ε, να υπάρχουν κανόνες ελέγχου, γιατί στηρίζουμε ανεπιφύλακτα το ελεύθερο εμπόριο στον τομέα αυτό με την Κολομβία και το Περού, όμως δεν θεωρούμε ότι πρέπει και άλλες χώρες να εκμεταλλευτούν από αυτή τη συμφωνία από την Κολομβία και το Περού. Στο γεωργικό τομέα υπήρξε και εκεί ε, δυναμική, θετική, στον τομέα των πνευματοδών ποτών. Ε, υπάρχει μια σημαντική συμφωνία με πολλά θετικά στοιχεία και όπως γνωρίζετε ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιεί σημαντικές διαπραγματεύσεις στον τομέα αυτό και σε διάφορες περιοχές. Τέλος, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών γνωρίζουμε ότι υπάρχει ε, σκληρός ανταγωνισμός στις αγορές αυτές από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Γι' αυτό λοιπόν εκτιμούμε ιδιαίτερα τις ε, προσπάθειες που καταβάλουν η Κολομβία, το Περού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις. Επιθυμούμε να βοηθήσουμε την επιτόπια βιομηχανία γιατί έτσι θα υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις και αυτό είναι το κλειδί της ανάπτυξης. Μίλησα λίγο και για τα συμφέροντα των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Θα μιλήσω ίσως για ευαίσθητα θέματα που αφορούν τη διακυβέρνηση, τα εργατικά δικαιώματα, τα ε, στοιχεία βιωσιμότητας που χαρακτηρίζουν τη συμφωνία. Ε, είπα από την αρχή ότι το πρόγραμμα Business Europe στηρίζει το σεβασμό και την εφαρμογή των δεσμεύσεων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ε, αλλά και άλλες διεθνείς ε, συνθήκες τις οποίες έχουν προσυπογράψει το Περού, η Κολομβία και άλλες χώρες. Αν δέχεται κανείς μια συμφωνία πρέπει και να την εφαρμόζει. Στηρίζουμε επίσης τα στοιχεία βιωσιμότητας που υπάρχουν σε αυτή τη συμφωνία κυρίως με το Περού και την Κολομβία. Κατά τη δική μας άποψη πρέπει να ε, συνεργαστούμε και με άλλους κοινωνικούς εταίρους, συνδικάτα, ε, κοινωνία των πολιτών, έτσι ώστε να δραστηριοποιήσουμε, να ενεργοποιήσουμε αυτό το στοιχείο της ε, βιωσιμότητας. Το στοιχείο της βιωσιμότητας είναι ένα νέο στοιχείο, θα είναι νέο για την Κολομβία, ήταν για το Περού, Μπορούμε λοιπόν να δεχτούμε την εφαρμογή αυτού του κεφαλαίου της συμφωνίας για να διασφαλίσουμε στοιχεία που αφορούν ε, στην εργασία και άλλα θέματα. Κάτι άλλο που θέλω να προβάλλω είναι το εξής. Εάν πρέπει να ληφθούν μέτρα για το εμπόριο, λόγω του ότι υπήρξε αποτυχία να εφαρμοστούν στοιχεία βιωσιμότητας, είτε αυτά αφορούν στο περιβάλλον, στην εργασία, είτε σε άλλους τομείς, επιθυμούμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβουλευτεί με τις οργανώσεις εργοδ εργοδοτών και εργαζομένων στην Κολομβία και το Περού πριν ληφθούν μέτρα. Ε, κατανοούμε υπάρχουν ε, ε, ομάδες που επιθυμούν να τοποθετηθούμε. Εμείς όμως ως οργάνωση των εργαδοτών θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξουν διαβουλεύσεις με τους φορείς που σας ανέφερα πριν ληφθούν περαιτέρω μέτρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Adrian. Πολύ ωραία απόψη χρόνου. Δίνω το λόγο στον κύριο Εδωάρδο Εστέβες, που είναι σύμβουλος ε, της Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε του Περού, κύριε Αντιπρόεδρε της Βολιβίας, προσκεκλημένοι, θα σας ευχαριστούμε που οργανώσατε αυτή την ακρόση. Θα ήθελα συνοπτικά να παρουσιάσω τις θέσεις την ε, Συνομοσπονδία Συνδικάτων της Αμερικής. Από την αρχή που άρχισαν ε, οι διαπραγματεύσεις είχαμε εκ μέσου όλων των συνδικάτων μεγάλες προσδοκίες για να δημιουργηθεί μια νέα σχέση και νέοι δεσμοί που θα συνδέουν όλες τις χώρες και όλους τους λαούς μας. Αυτά τα δέκα χρόνια συνεργασίας και διαλόγου πολιτικού πιστεύουμε ότι ακόμη δεν έχει εξευρεθεί το κατάλληλο ισορροπημένο πρότυπο. Στα πλαίσια των συνδικαλιστικών μας δράσεως προτείναμε η συνδικαλιστική σχέση μεταξύ ημών και ημών να διευρυνθεί για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε θέματα μετανάστευσης και κοινωνικοεργασιακά. Σήμερα μας ανησυχεί το γεγονός ότι η συνθήκη την οποία εξετάζουμε έχει πάρα πολύ ισχυρό σκέλος εμπορικό και λιγότερο αναφέρεται στα θέματα τα οποία αφοράν τις υπηρεσίες. Στα πλαίσια των ε, συντονιστικών οργάνων μας κάναμε έκκληση Μήπως μπορείτε να τρέχετε λιγότερο, λέει ο πρόεδρος, για να καταλάβουμε και εμείς τι λέτε. Δώστε μου άλλο ένα λεπτό και θα μιλήσω. Πιο αργά. Λοιπόν, το 2010 όλες οι οργανώσεις που προανέφερα Κάναμε έκκληση στις κυβερνήσεις μας κατά τη διάρκεια της ασκέψης κορυφής της Μαδρίτης και ζητήσαμε να μην υπογραφούν οι συμφωνίες με την Κολομβία και το Περού, δεδομένου ότι θεωρούμε ότι είναι αντιφατικές σε σχέση με την ενδυνάμωση που θέλαμε, δεδομένου ότι πρόκειται μόνο για μια συνθήκη ελευθέρου εμπορίου και δεν λαμβάνει υπόψη τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, κυρίως τη βία που υπάρχει στην κοινωνία της Κολομβίας. Επίσης, ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν διάφοροι κινδυνοί που υφέρπουν και δεν ζητούμε να επικυρωθεί η συμφωνία αυτή. Για ποιους λόγους. Πρώτα απ' όλα, θέλουμε να αναδιορθωθεί η συζήτηση για την ανάπτυξη και να πούμε ότι θέλουμε να αναπτυχθεί η παραγωγή, να ληφθούν υπόψη τα περιβαλλοντικά θέματα η φόρος ανάπτυξη, η αύξηση των εισοδημάτων, η βελτίωση της ασφάλειας στην εργασία, η ποιότητα ζωής. Στην προηγούμενη περίοδο κατά την οποία μελετήθηκε αυτή η συνθήκη, πρέπει να πω ότι όλα αυτά τα θέματα μας τα είχαν αρνηθεί. Γίνεται συσσόρευση ε, των χρεών του ΙΔΑ και πλουτισμός ολίγων. Θέλουμε να αλλάξουν τα πράγματα. Η συμφωνία αυτή θα πρέπει να δώσει περισσότερη δύναμη σε τις οργανώσεις των εργαζομένων και θα θέλαμε ε, η εξουσία η οποία δίδεται στις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις να μπορέσει να μειωθεί μέσω συμφωνιών. Επίσης, το θέμα της περιφερειακής και δημερού συνεργασίας είναι ένα θέμα το οποίο έχει φύγει από τη μέση με τη συμφωνία αυτή. Και εμείς θα θέλαμε η συνεργασία σύνταξη όλων των χωρών να γίνουν ώστε να μπορέσει να υπάρχει συντονισμένος διάλογος, συνεργασία και διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες εμπορικών σχέσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μας στα πλαίσια της ανάπτυξής μας. Και η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να μας βοηθά να αναπτυχθούμε περισσότερο. Αυτά όμως τα θέματα αφέθηκαν στο περιθώριο και γι' αυτό είμαστε εναντίον αυτή τη συμφωνίας. Επίσης θα πρέπει να πω ότι δεν λύνεται επίσης το πρόβλημα της συνδικαλιστικής βίας την οποία αντιμετωπίζουμε στην Κολομβία. Οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν τα τελευταία χρόνια για μεταξύ των ε, εργαζομένων ε, και των, ε, της κυβέρνησης η ποινικοποίηση καταστρατήγησης των συνδικαλιστικών δράσεων και άλλα θέματα είναι μια κάποια βελτίωση της κατάστασης, αλλά υπάρχουν ακόμη εκρεμή και άλλοι πάρα πολλά θέματα τα οποία μας αφορούν. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει τέτοιου είδους καταστάσεις να επαναλαμβάνονται και αν δεν υπάρξει ε, δράση εκ μέρους της κυβέρνησης ώστε να σταματήσει η ατιμορρησία των δολοφονιών κατά των ε, καλλιτικών οργάνων δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Υπάρχουν τελευταία νέα τα οποία δεν μπορούσα ακόμη να αναλύσω για να σας πω αν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η ευελιξία των συνθήκων εργασίων, η καταστρατήριση των δικαλιστικών δικαιωμάτων και σιγά σιγά η καταστροφή των συνδικάτων δεν είναι κάτι που μας βρίσκει σύμφωνους. Πάντα υπάρχει η απειλή των ενεργειών του ανθρώπου στο περιβάλλον. Και το δραματικό πρόβλημα που δημιουργείται για όλους από την ε, κλιματολογικές αλλαγές είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Επίσης, ε, αναφέρομαι κυρίως σε δραστηριότητες της εξωτερικής, βιομηχανίας, άλλες δραστηριότητες τις οποίες είναι όλο και περισσότερο εντατική η εργασία και στην οποία απασχολούνται όλο και λιγότερα άτομα. Πρέπει να πω ότι πάρα πολύ μεγάλα μέρη του πληθυσμού αυτόχθονες και άλλοι με τις δραστηριότητες τους δημιουργούν προβλήματα στην, ε, στο περιβάλλον μας ε, και στην ισορροπία μας. Όλο και περισσότερο οι χώρες μας θα συνεχίσουν να ε, προσφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντα τα οποία οδηγούν στην σπάνη και στην εξασθένηση των πλουτοπαραγωγικών φυσικών μανπόρων χωρίς να υπάρχει καμία αντι, κανένα αντιστάθμισμα. Αυτά τα μεγάλα προϊόν, ε, προβλήματα τα οποία υπάρχουν είναι προβλήματα που πιέζουν όλοι μας την κοινωνία. Θα ήθελα όμως να μας εξηγήσει η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση τι εννοεί σοβαρή καταστρατήγηση των δικαιωμάτων και νομίζω ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει και να συμφωνηθεί στα πλαίσια της συμφωνίας αν δεν έρθει σε επαφή με τους κοινωνικούς εταίρους. Ξέρουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν ε, στην παρούσα ε, κατάσταση αλλαγές στην και Γι' αυτό ζητούμε να μην υπογραφεί. Κατά την άποψή μας θα πρέπει αυτές οι εμπορικές συμφωνίες να θεωρηθούν ως προσωρινές συμφωνίες για τις οποίες αρκεί μόνο η επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο του Πρόεδρου δεδομένου ότι η Κολομβία δεν χρειάζεται επικύρωση. Ε, επειδή έχω πάρα πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μου, αν θέλετε, το, η γραπτή μου ομιλία είναι στη διάθεσή μας. Ο χρόνος είναι ίδιος για όλους, λέει ο Πρόεδρος. Ε, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Σας έδωσα για μισή λεπτό παραπάνω από αυτό που προβλεπόταν. Περνούμε στον κύριο Οράσιο Γουίντο από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας που εκπροσωπεί την κυρία Κλεοπάτρα Ντομιά Χέρινγκ. Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του ILO. Πού κάθεστε? Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Επιτροπή, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρα της Βολιβίας, κύριε Αντιπρόεδρε του παιδού, κύριε και κύριοι συμμετέχοντε, σας ευχαριστώ που καλέσατε τον ΔΟΕ, που όλο και περισσότερο βλέπει σε όλες τις εμπορικέ διμερεί και περιφερειακές συμβολίε να συμπεριλαμβάνονται τι δύο τελευταίε δεκαετία ρήτρε που αφορούν τι εργασιακέ σχέσει και θα πρέπει να ευρεθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί ώστε να εφαρμοστούν σωστά οι κανόνες που μας διέπουν. Θα πρέπει να τονίσω ότι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα αν θα πρέπει ναι ή όχι να υπογραφεί μία εμπορική συμφωνία με μία τρίτη χώρα, διότι είναι θέμα δική του κυριαρχία. Παρ' όλα αυτά, οποιαδήποτε η πρωτοβουλία έχει σχέση με τι διεθνεί κανόνε εργασία του ΔΟΕ είναι καλοδεχούμενη η δήλωση του ΔΟΕ για την ε, κοινωνική δικαιοσύνη στα πλαίσια της ε, διακήρυξης του 2008 έχει ως στόχο να παρέχει βοήθεια στα μέλη τα οποία θέλουν να προωθήσουν συλλογικά τους στρατηγικούς στόχους στα πλαίσια διμερών ή πολυμερών συμφωνιών όταν συνάδουν με τις ε, συμβάσεις που έχουν σε σχέση με τις αρχές του ΔΕΔΕ. Όσον αφορά τις εργασιακές ρήτρες, τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα σχετικές εκθέσεις που έχουμε εμείς βάσει των ε, εκθέσεων των εμπειρογνωμόνων, των ε, επιτροπών ad hoc και ιδιαίτερως τις συστήσεις της ε, Επιτροπής Συνδικαλιστικής Ελευθερίας του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Επίσης, πρέπει να πω ότι ε, αυτές οι συμφωνίες εφαρμόζονται σε αυτούς που δεν έχουν ε, συνάψει τις ρήτες. Και βεβαίως οι πάντες μπορούν να συμβουλευθούν τις εκθέσεις που υπάρχουν ε, εκ μέρους των οργάνων εποπτείας. Τα σχόλια και τα μέτρα που κάνουν οι κυβερνήσεις και τα μέτρα τα οποία υιοθετούν είναι κάτι το οποίο μας επιτρέπει κάθε φορά να προχωρήσουμε. Θα αναφερθώ, επειδή έχω πάρα πολύ λίγο χρόνο, σε θέματα, τα κύρια θέματα, τα οποία τονίστηκαν ως ε, εμπόδιο για την ε, άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Το κύριο πρόβλημα το οποίο εντόπισε για την άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων ε, και ανέφερε η Κολομβία είναι το θέμα της βίας κατά των συνδικαλιστικών ορών και μέσω μηχανισμών και αποστολών προσπαθούμε να ερευνήσουμε την κατάσταση και βλέπουμε ποιες είναι οι σχετικές διατάξεις. Πρέπει να πω ότι με τις εκθέσεις ε, των ε, οργάνων εποπτείας και με τις διάφορες διάφορα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι διάφορε αποστολές ε, είδαμε ότι υπήρχαν τέτοιου είδους επιπτώσεις. Είδαμε παρόλα αυτά ότι αναγνωρίζεται το δικαίωμα διαπραγμάτευσης για συλλογική ε, δια, ε, σύμβαση στον δημόσιο τομέα και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε το πρόβλημα της, στο πρόβλημα της βίας κατά των συνδικαλιστικών οργάνων βλέπουμε ότι έχουν υπάρξει μέχρι τώρα 250 δολοφονίες συνδικαλιστικών οργάνων. Επίσης έχουμε δει ότι υπάρχουν διάφορες δράσεις εκ μέρους ε, των ε, υπευθύνων και των κυβερνήσεων ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν προστατευτικά μέρα και να η βία κατά των συνδικαλιστικών οργάνων. Έτσι, από πέρσι, το 2000, ε, από το Φεβρουάριο του 2010 μέχρι σήμερα, έχει πέσει σε 48 ε, ο αριθμός των συνδικαλιστών που έχουν δολοφονηθεί. Ξέρουμε ότι πρόκειται για θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ τον Τρία τελευταία χρόνια η Επιτροπή Υπηρογνωμόνων διαπίστωσε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση των κονδυλίων τα οποία δίδονται στα ερευνητικά όργανα για να ερευνήσουν την κατάσταση και έχουν ε, ληφθεί και δικαστικές αποφάσεις και καταδικαστικές αποφάσεις κατά αυτών οι οποίοι ε, δολοφονούν συνδικαλιστές. Ξέρουμε ότι τους τελευταίο 1,5 χρόνο έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των καταδικαστικών αποφάσεων κατά αυτών των ατόμων που θεωρήθηκαν ένοχα. Παρ' όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί, όπως είπα προηγουμένως, ο αριθμός των δολοφονιών, θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να σταματήσουν αυτές οι δολοφονίες ε, οι οποίες άρχισαν τη δεκαετία του 80 και θα προσπαθήσουμε μέσω δικαστικών ή εξοδικαστικών οδών να διευκρινίσουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει να πω ότι τις σχετικές ε, συμφωνίες τις έχει επικυρώσει. Όσον αφορά την συγκεκριστική ελευθερία βάσει της ε, Σύμβασης 87 του Περού, κάνουμε εμείς ε, διάφορες παρατηρήσεις για το δικαίωμα συνδικαλιστικής, ε, ανάπτυξης συνδικαλιστικής δράσης, το δικαίωμα απεργίας και άλλα θέματα τα οποία αφορούν τους εργαζόμενους και ζητήσαμε από την κυβέρνηση να λάβει τα σχετικά νομοθετικά μέτρα και να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις ώστε οι επόμενες ε, συλλογικές ε, συμβάσεις να λαμβάνουν υπόψη, κυρίως 87 και 94, να λαμβάνουν ε, υπόψη τα δικαιώματα των εργαζομένων, των συνδικαλιστών και να προβλέπουν τα κατάλληλα μέτρα και τις κυρώσεις. Επίσης, πρέπει να πω ότι υπάρχουν ε, σχετικοί νόμοι που αφορούν τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα καθώς και εμπόδια τα οποία τίθενται για την άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων. Θα σας διαθέσω για τη γραπτή μου έκθεση για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στον Επίτροπο Ντεχούχτ, μπορώ να σας πω ότι όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα θα βρίσκονται στη διάθεση των μελών της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ. Επίτροπε σας καλωσορίζω και πάλι. Έχετε συνηθίσει βεβαίως ε, να μιλάτε εδώ. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε και κυρία Αντιπρόεδρε, ε, αξιότιμα μέλη Χαίρομαι πολύ για την ε, δυνατότητα που έχουμε να συζητήσουμε εδώ τη Συμφωνία Εμπορίου ε, με το, Περού και την Κολομβία. Είναι πολύ σημαντική συμφωνία για όλα τα ενδιαφέρομενα μέρη που θα βοηθήσει την, στην ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων. Για την Κολομβία και το Περού αυτή η συμφωνία θα βελτιώσει και θα διευκολύνει την, ε, την πορεία τους προς την οικονομική ευημερία και την ανάπτυξη. Για την Ευρώπη η συμφωνία αυτή είναι άλλο ένα βήμα ε, και ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να βγούμε από την δύσκολη οικονομική συγκυρία που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Πρώτα για τον οικονομικό αντίκτυπο της, ε, της ε, συμφωνίας. Όταν εφαρμοστεί πλήρως θα υπάρχουν σημαντικά ωφέλη σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη. Θα ενισχύσει την ανάπτυξη των εταίρων μας κατά 1% του ΑΕΠ και σε γενικές γραμμές ε, περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ θα εξοικονομούνται κάθε χρόνο μόνο και μόνο από δασμούς, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε 100% τερματισμό των ε, ε, τελωνιακών ελέγχων σε αρκετούς τομείς το Περού και η Κολομβία θα ε, απομακρύνουν όλους ε, τους δασμούς ε, μετά από το τέλος μιας δεκαετούς μεταβατικής περίοδου. Και έτσι οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς θα ξεκονομήσουν τουλάχιστον 250 εκατομμύρια ευρώ κατά έτος σε δασμούς. Για να σας το πω πιο ξεκάθαρα, 60 από την κλωστεφαντουργία, 30 από την αυτοκινητοβιομηχανία, 10 εκατομμύρια για τα αλκοολούχα ενοπνευματόδη ποτά και 18 για τις τηλεπικοινωνίες. Από την άλλη υπάρχουν και ε, προοπτικές για ανάπτυξη με την, ε, τις ανεξάρτητες μελέτες που θα αυξήσουν τον, το ΑΕΠ κατά 0,7 και 1% αντίστοιχα. Οι εξοικονομήσει σε δασμού θα ε, ανέρχεται σε πάνω από 50 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Επιπλέον θα υπάρχει και μια σειρά ε, λιγότερο απτών αλλά εξίσου σημαντικών οικονομικών ε, επιπτώσεων. Ε, νέες οικονομικές και επενδυτικές δυνατότητες, μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας που αυξάνει τη δυνατότητα για την ανάπτυξη της οικονομίας, την κοινωνική συνοχή και την ισότητα ευκαιριών. Πράσινη ανάπτυξη επίσης άλλη πολύ σημαντική πτυχή, αλλά και ίση όρια ανταγωνισμού σε όλες τους τομείς ε, της αγοράς και στι δημόσιε προμήθειες, τα πνευματικά δικαιώματα και ούτω καθεξής. Η συμφωνία μετά έχει και, ένα συνδυασμό αυτών των συστημικών ε, ε, επιπτώσεων σε ένα κοινό σύνολο κανόνων που θα ενισχύσουν την εταιρική σχέση των περιφερειών μας μια εταιρική σχέση που θα σταθεί στο ύψο ε, όλων των προκλήσεων που ενδεχομένω να αντιμετωπίσουμε τον 21ο αιώνα. Όμω, εδώ δεν μιλάμε μόνο για business, γιατί η επιχειρηματική δράση έχει αντίκτυπο και στην κοινωνία και πρέπει να το φροντίσουμε και αυτή την τυχή. Τμήμα της, ε, του σημερινού διαλόγου αφορά τον ρόλο της ε, ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής και πώς επηρεάζει και την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που έχω πει επανειλημμένα ενώπιόν σας ε, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την Κολομβία και το Περού. Αυτή η συμφωνία θα στηρίξει τις, ε, την κοινωνική συνοχή ε, της Κολομβίας και του Περού που είναι θεμελιώδη στοιχείο για την ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Και για την αηφόρα ανάπτυξη βεβαίως αν η Ευρώπη απομακρυνθεί από μια τέτοια συμφωνία, θα αμελούσε όλα αυτά τα καθήκοντα που έχει και τι δεσμεύσει που έχει αναλάβει, θα αφήσει την Κολομβία και το Περού σε ένα... και θα χάσουν έτσι αυτές οι δύο χώρες την ευκαιρία από ένα βίο παρελθόν να πάνε σε μια δημοκρατική κοινωνία στο μέλλον. Βεβαίως πρέπει να προσέξουμε την ε, διασφάλιση των δημοκρατικών και συνεκολαστικών δικαιωμάτων και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να στηρίξουν τη συμφωνία για αυτού τους λόγους. Θα ήθελα να πω ότι και εγώ συμμερίζομαι την επιθυμία σα ε, να προωθήσουμε τα, όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και των συνδικαλιστικών και ξέρω ότι ο πρόεδρο Σάντο θέλει να το κάνει αυτό. Ε, Όπω και ο πρόεδρο Γανζόν. Εγώ είμαι απολύτω πεπισμένο ότι η συγκεκριμένη εμπορική συμφωνία με, τα κίνητρα που παρέχει θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ε, κοινωνία των πολιτών της Κολομβίας ε, και την κατάσταση ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό όχι μόνο στην Κολομβία, αλλά και σε όλε τι χώρε που ε, ε, αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Σε αυτέ τι χώρε, λοιπόν, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι αιτίε του προβλήματο, δηλαδή η ακραία φτώχεια και ο κοινωνικό αποκλεισμό. Ο καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα είναι η συνεκτική οικονομική ανάπτυξη. Ε, καταβάλουμε λοιπόν ε, προσπάθειες ε, για να ενισχύσουμε τη συνεργασία, να μειώσουμε την φτώχεια και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Ε, ως εκ τούτου θα έχει άμεσο αντίκτυπο και στα ζητήματα της δημοκρατίας και τη δικαιοσύνη. Όπως είπαν και οι αντιπρόεδροι Κρούς και Καζόν και σίγουρα θα το επιβεβαιώσουν, αυτή η συμφωνία δεν είναι μόνο ισχυρή στι αρχέ τη, αλλά εύρωστη και σε ό,τι αφορά τι νομικέ της δεσμεύσει εξασφαλίσαμε ότι αυτές οι αρχές που συμφωνήσαμε να προωθήσουμε καταγράφονται και στι διατάξεις και ε, θα διατρέξω τις διατάξεις που, είναι, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρώτον, οι διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που διασκεδάζουν τις ανησυχίε σας για τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα. και θα λαμβάνουν υπόψη και τον, ευρύτερο ευρωπαϊκό στόχο για την ε, διασφάλιση του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών ελευθεριών. Δημοκρατικές ελευθερίες λοιπόν, ε, στο άρθρο 1 συμπεριλαμβάνονται ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι δημοκρατικές ελευθερίες, εργασιακές ελευθερίες, όλα αυτά που βασικά στοιχεία της συμφωνίας. Αυτό σημαίνει ότι, ότι αν μια κυβέρνηση παραβιάσει αυτά τα βασικά στοιχεία, τα άλλα μέρη θα είναι σε θέση αμέσως και μονομερός να άρουν ε, τα ωφέλη της, ε, και να ανακαλέσουν τα ωφέλη της συμφωνίας στα άλλα μέρη. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να εκφράσουμε κάτι τέτοιο με πιο ισχυρό τρόπο και πιο ξεκάθαρο τρόπο. Ξέρω ότι έχετε ανησυχίε σε ό,τι αφορά τι εσωτερικέ ε, διαδικασίε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να οδηγήσουν σε αυτή την ανάκληση. Όμω, εγώ δεσμεύομαι ότι θα εφαρμοστούν με πολύ σοβαρό τρόπο αυτέ οι συμφωνίε. Και αυτό είναι με εξίσου σοβαρό τρόπο όσο για, για τις υπόλοιπες οικονομικές ε, διατάξεις. Ο θεμιόλιος μας στόχος ε, να ε, εξηγειάνουμε και να ενισχύσουμε την, τις δημοκρατικές ελευθερίες θα είναι ο κύριος μας στόχος. Ενώ διατηρούν την εθνική τους κυριαρχία. Τα, κράτη τα, τα μέρη μάλλον της συμφωνίας ε, συμφωνούν ε, να τηρήσουν ε, τους στόχους για τους όρους της συμφωνίας και να εφαρμόσουν τις οκτώ κύριες συμβάσεις του ΔΟΕ και τις κύριες περιβαλλοντικές συμφωνίες. Υπάρχουν, και υπάρχει συγκεκριμένος μηχανισμός επίλυσης διαφορών ο οποίο μπορεί να κινηθεί από οποιοδήποτε μέρο, ακόμα και αν διαφωνούν τα υπόλοιπα μέρη. Η διαδικασία γίνεται από ανεξάρτητους ε, και αντικειμενικούς ε, εμπειρογνώμονες ε, και βάσει αυτού του μηχανισμού μπορεί να ληφθεί άμεση απόφαση και εφαρμογή αυτής της απόφασης. Ε, θα υπάρχουν βεβαίω και ομάδε κοινωνία των πολιτών σε κάθε μέρο, συμβαλλόμενο μέρο. Ε, και εμεί βασιζόμαστε στην ενεργό του ε, συμμετοχή για να μπορούν να επιστούν την προσοχή μα σε συγκεκριμένα προβλήματα. Για παράδειγμα, θα υπάρχουν ανοιχτέ συνεδριάσει ε, των διοικητικών θεσμών, όπου οι πολίτε και οι κοινωνία των πολιτών θα μπορούν να γύρουν ζητήματα. και όλες οι αποφάσεις θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Με όλε αυτές τι δικλείδες ασφαλεία. μπορείτε να συμφωνήσετε μαζί μου ότι ε, η συμφωνία αυτή είναι, ε, θα διασφαλίζει την ε, τήρηση και τον σεβασμό των δημοκρατικών ελευθεριών. Θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, Πρόεδρε, ακόμα να την υιοθετήσουμε και φέτος το καλοκαίρι και πάλι θα πρέπει να υιοθετηθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Κάτι μπορεί να γίνει σύντομα, αν το επιθυμούμε. Εγώ προσωπικά ελπίζω να τεθεί σε ισχύ το στομότερο δυνατόν, γιατί είναι ε, σημείο κλειδί στη στρατηγική μα για την οικονομική ανάπτυξη τη περιφέρεια και ε, πληρεί του όρου που έχουμε θέσει σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αηφόρα ανάπτυξη. Προσβλέπω σε συνεργασία μαζί σα και σα ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. <clears throat> Commissioner. Let's move to Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Θα ας προχωρήσουμε τώρα. Τους προσκεκλημένους μας από την Κολομβία και το Περού ξεκινάω με τον Αντιπρόεδρο Αγγελίνο Καρτάν από την Κολομβία. Και θα ήθελα επίση ε, να σας πω ότι έχουμε κοντά μας ε, και επίσημη εκπροσώπηση από αυτή τη χώρα τον κύριο Σιμών Καβίρια, ο οποίος είναι πρόεδρος ε, της ε, Βουλής των Αντιπροσώπων, της Κάτω Βουλής αν θέλετε, της ε, Κολομβίας. Και έχουμε και τον ηγέτη, τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος. Και αν μας μείνει λίγος χρόνος θα τους δώσω το λόγο για σύντομη παρέμβαση, αλλά δεν σας το υπόσχομαι. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Αντιπρόεδρο για 10 λεπτά παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω με όλο το συμβασμό το εξή. Δεδομένου ότι έχουμε μαζί μας την Αντιπρόεδρο του Περού, την κυρία Μαρισόλε Σπινόσα Κρούθ, και για να ποτίσουμε φόρο τιμή στις γυναίκες προέδρους της Λατινικής Αμερικής, της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της Πρωθυπουργού της ε, να δώσουμε πρώτα το λόγο στην εξαιρετική πρώτη αντιπρόεδρο του Πυρού, την κυρία Μαρισόλ Εσπινός Ακρούς. Ακολουθώ την υπόδειξή σας και θα δώσω πρώτα το λόγο στην ε, πρώτη αντιπρόεδρο του Περού, την κυρία Μαρισόλε Σπινόσα Κρούτ. Να σας πω επίσης ε, ότι υπάρχει και μία πολύ άριθμη αντιπροσωπή από το Περού που αποτελείται από τον Χωσέ Λουί Σίλβα, ο οποίος είναι υπουργό Εμπορίου και Τουρισμού, τον κύριο Μανουέλ Μπουλγκάρ Πιδάλ, υπουργό ε, Περιβάλλοντος, κύριος Εντουάρντο Μπραντές, Εθνικός Διευθυντής των Διεθνών Διαπραγματεύσεων Εμπορίου και Τουρισμού και τον πρέσβη Φερνάντο Ρόχας, που είναι Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Σας καλωσορίζουμε όλους σας θερμά. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα τον την Αντιπρόεδρο από το Περού. Για 10 λεπτά παρακαλώ. Μαρίσες Πινάσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αποφθύνω χαιρετισμό σε εσά κύριε Πρόεδρο Βιτάλ Μορέλ, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Εκνοβίου, να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου Αγγελίνο Γαρθών που είναι υπότης να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Καρέλ Ντεκούρχ, υπεύθυνο για το εμπόριο. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, σήμερα στην αντιπροσωπεία μου με, αντιπροσωπε... με... συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικού Εμπειρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και μία αντιπροσωπεία από την πρεσβεία μας, πράγμα το οποίο επικυρώνει την βούλησή μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω στη δυνατότητα που δίδεται στη χώρα μου να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε αυτή την δημόσια ακρόαση, να σας απευθύνω τον χαιρετισμό του Προέδρου μας Μαλατάσο και να σας τονίσω πόσο σημαντική είναι η συμφωνία αυτή για τη χώρα μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για μας είναι ένας από τους πιο σημαντικούς εμπορικούς εταίρους. Υπό ποια έννοια όχι μόνο είμαστε από ιστορικής πλευράς συνδεδεμένοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όλο και περισσότερο μέσα στο χρόνο ενισχύονται όχι οι δεσμοί συνεργασίας, αλλά και ο... οι προσπάθειες ενίσχυσης της ε, δημοκρατίας στη χώρα μας, δεδομένου ότι έχετε στείλει αντιπροσωπείες παρατηρητών ε, όταν έχουμε εκλογές και μας έχετε βοηθήσει για την παγίωση των ανθρωπίνων και συνδικαλιστικών ε, δικαιωμάτων. Το Περού είναι μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία της οποίας η μακροπολιτική ε, οικονομική πολιτική βασίζεται σε σταθερότητα και θέλει με τα προγράμματά της να μπορέσει να καταπολεμήσει την φτώχεια, να θεσπίσει συνθήκες σωστής εργασίας και να βελτιώσει τους στόχους της χιλιετίας. Ένας από τους αντικειμενικούς στόχους προτεραιότητας είναι η κοινωνική ανάπτυξη και η οικονομική ανάπτυξη που θα μας βοηθήσουν όχι μόνο να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, αλλά να μας επιτρέψει σε όλους σε εμάς και σε όλους τους μικρούς παραγωγούς να σταματήσουν να είναι αόρατοι πολίτες, αλλά να γίνουν συντελεστές οικονομικής ανάπτυξης χώρες μας. Γι' αυτό θέλουμε να υπάρχει για τον εμπορικό κόσμο ένα κτήμα θετικό, θέλουμε να υπάρξει άνοιγμα προς τις επενδύσεις και αυτό να μπορέσει να αγκαλιάσει όλους τους τομείς της οικονομίας και όλες τις περιοχές όχι μόνο την περιοχές της παράκτιες, αλλά και τις ορεινές, ημιορεινές και άλλες φτωχές περιοχές. Για να μπορέσουμε λοιπόν ε, να κάνουμε πραγματικότητα τις υποσχέσεις μας, το 20% των πόρων μας ε, έχει δοθεί για την προάστηση κοινωνικών θεμάτων για να βελτιωθεί η κοινωνική πολιτική, η υγεία και η εκπαίδευση. Δημιουργήθηκε ένα ειδικό Υπουργείο και αυτή τη στιγμή κάνουμε πολιτικές δεύτερης γενιάς, διότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε όχι μόνο τη φτώχεια, αλλά θέλουμε να βγουν από αυτό το κλίμα φτώχεια οι άνθρωποι και να μπορέσουν να αποτελέσουν μέρος του παραγωγικού μας ιστού. Πρέπει να πω ότι το 2016 θέλουμε να έχουμε μόνο 3 εκατομμύρια Περουβιανούς που ζουν κάτω από ε, το κατόφλι της στόχιας, δηλαδή λιγότερο από 20% έως το 2016 και γι' αυτό προσπαθούμε να ενεργήσουμε σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Τα... Η εμπορική αυτή συνωνία, συμφωνία θα είναι μια εξαιρετική συμφωνία κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους μικρομεσαίους παραγωγούς και για τα άτομα τα οποία ζουν στην Ήπεθρο, διότι αποτελούν το 98% των επιχειρήσεων και 95% του πληθυσμού μας. Εμείς ε, είμαστε μάρτυρες και εγώ ως εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου, εκτός από αντιπρόεδρος, είμαι μάρτυρας του πώς η παραγωγή, και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικονομική συνεργασία μας Ένωση και κυρίως να ευχαριστήσω τους Γερμανούς, τους Γάλλους, τους Ιταλούς που άρχισαν να ανοίγουν τις πόρτες τους ε, εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες και άρχισαν να συνεργάζονται με τους μικρούς παραγωγούς καφέ και κακάο. Εγώ είμαι μάρτυρας αυτής της πείρας, ότι αν ένας παραγωγός με τεχνολογία, με συνεργασία, αλλά κυρίως εάν του ανοίξουν τις πόρτες οι διεθνείς αγορές είναι όχι μόνο σε θέση να βγει από τη φτώχεια αλλά να κάνει ακόμη ένα βήμα προς τα μπρος και αυτοί είναι ο στόχος κυβέρνησής μας. Θέλουμε επίσης κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές να τονίσουμε την δέσμευση που έχει ο πρόεδρος Ουμάλα για την διασφάλιση του περιβάλλοντος. Έχουμε με το θέμα των εξορυκτικών βιομηχανιών μας ε, νέες ιδέες που θα σέβεται δύο βασικές παραμέτρους. Πρώτα απ' όλα έχουμε το θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων και το δεύτερο, η δεύτερη παράμετρος είναι το θέμα της στήρησης και σεβασμού του περιβάλλοντος, διότι αυτό κάποια χώρα η οποία θέλει να επιτύχει αηφόρο ανάπτυξη, δεν θα μπορέσει να Όποια χώρα θέλει να επιτύχει αηφόρο ανάπτυξη, δεν μπορέσει να κάνει τίποτε εάν δεν λάβει υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό για μας είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Επίσης, η αλλαγή των προτήτων παραγωγής και κατανάλωσης είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επίσης, θέλουμε αυτή τη δέσμευση ε, για μία εξορρυκτική βιομηχανία υπεύθυνη, να την επαναλάβουμε. Ο πρόεδρος Ουμάλα θέλει να έχουμε μία διαφορετική πολιτική και έχουμε νέους νόμους που ε, αφορούν και τα θέματα της ε, φορολογίας. Επίσης, πρέπει να πω ότι ο πρόεδρος μας προσέχει ιδιαίτερα την ε, σεβασμό και την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Αυτό που μας απασχολεί είναι να γίνουμε πραγματικά ένα κράτος δικαίου που θα είναι σε θέση να σέβεται ακόμη και αυτές τις τελευταίες ε, εβδομάδες που συλλάβαμε την, ε, τον αρχηγό μίας τρομοκρατικής οργάνωσης, ακόμη και αυτού να του εξασφαλίσουμε την κατάλληλη υπεράσπιση των δικαιώματών του. Έχουμε επικυρώσει επίσης τα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών τη Σύμβαση, τη σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και επίσης ε, έχουμε σε θέματα εργασιακά, όπως είπε και ο εκπρόσωπος ε, της Διεθνής Οργάνωσης Ιδία τις 67 σχετικές συμβάσεις. Το θέμα του διαλόγου το ενισχύουμε, τα εργασιακά δικαιώματα τα βελτιώνουμε και το δικαίωμα του συνέρχεστε επίσης το τηρούμε. Θέλουμε να γίνονται σεβαστά επίσης τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, να προσθεθούν στα ανθρώπινα δικαιώματα και θα εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Η συμφωνία αυτή είναι διαφορετική από άλλες τις οποίες έχουμε υπογράψει. Διότι δεν είναι μόνο εμπορική συμφωνία, αλλά συμπεριλαμβάνει και δύο ρήτρε. Η μία αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα, θα προσπαθήσουμε να υπάρχει συμμετοχή και δέσμευση με πνεύμα διαφάνειας και όλα αυτά να γίνουν με την επικύρωση της Βουλής μας. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που μας απασχολεί στην κυβέρνησή μας και έχουμε αναλάβει την δέσμευση να φέρουμε σε πέρα στο θέμα αυτό. Τώρα, όσον αφορά τις κοινότητες των αυτοκτόνων, πρέπει να πω ότι εμείς έχουμε προβλέψει ένα, μια ρήτρα πρώτερης διαβούλευσης ε, και προβλέπουμε κανονισμούς βάσει των οποίων προβλέπεται η συμμετοχή των διαφόρων κοινοτήτων στην οποία συμμετέχουν οι σχετικοί ε, φορείς και εκπρόσωποι όλων των διαφορετικών ε, κοινοτήτων αυτοχθόνων που υπάρχουν στη χώρα μας. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση στην οποία οι εκπρόσωποι των ε, πρώτων ε, κοινοτήτων αυτοχθόνων που ζούσαν στη χώρα μας να συμμετέχουν σε όλες τις συζητήσει που κάνουμε για βελτίωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την χώρα μας το θέμα της ε, πολυπολιτισμικότητας και της βιολογικής ποικιλομορφίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας και οι διαφορετικοί ε, σκηνότητες και άνθρωποι που ζουν στη χώρα μας εμπλουτίζουν τη χώρα μας. Επίσης καταβάλουμε προσπάθειες για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία των ε, εμπόρων ναρκωτικών. Η βούληση της κυβέρνησής μας είναι να πολεμήσουμε αυτούς τους τρομοκράτες. Και ο πρόεδρος του Μάλα το επιβεβαίωσε αυτό με την ε, σύλληψη του τελευταίου τρομοκράτη του Σεντέρο Λουμινόσο. Η πόλεμος κατά των ναρκωτικών είναι ένα θέμα το οποίο συμμερίζονται όλες οι χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κολομβία και το Περού. Θέλω να τονίσω ότι βρισκόμαστε σε διαδικασία αλλαγής σε διαδικασία ανάπτυξης μιας νέας κυβέρνησης που δίδει την δέουσα σημασία στο ανθρώπινο «ον» και κάνει ανθρωποκεντρική πολιτική. Θέλω επίσης να μιλήσω για μια χώρα, για ένα Περού για όλους. Ένα Περού που θα είναι το Περού της συμπερίληψης και όχι των αποκλεισμών. Θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη, αλλά η ανάπτυξη να γίνει με προστασία των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αηφόρων άπτυξης. Και ελπίζουμε ότι μπορούμε να υπολογίζουμε στην δική σας συνεργασία κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην οδό της ανάπτυξης που περιμένουν τόσο πολύ όλοι οι πολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα λοιπόν ε, ας ακούσουμε την ε, Αντιπρόεδρο Αγγελίν ε, τον Αντιπρόεδρο Αγγελίν Βαχιάν από την Κολομβία. Δέκα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε του Περού, κυρία Μαρισόλε Σπινόσα, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κοινωνίας των πολιτών και εκπρόσωποι της κοινωνίας μας του Περού και της Κολομβίας το Μάιο του 2010 η Κολομβία υπέγραψε τη εμπορική συμφωνία μεταξύ Κολομβίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κατόρθωσε η Βουλή μας να την εγκρίνει. Αυτή τη στιγμή ενεργούμε ώστε στα διάφορα επίπεδα και στους διάφορους θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επικυρωθεί αυτή η συμφωνία. Δεν έχουμε να κάνουμε με μια χάρη που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κολομβία. Ούτε με μια κατάσταση την οποία κάνει χάρη η Κολομβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια ισομερή συμφωνία. Για μια οικονομικά υποφελή συμφωνία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Κολομβία που συνεισφέρει στην πολιτική απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην πολιτική απασχόλησης και της Κολομβίας. Και όταν εμείς αποφασίσαμε να συνάψουμε και να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία, το κάναμε διότι ως πολιτικοί στη χώρα μας Θέλουμε η Κολομβία να γίνει μία χώρα που προοδεύει. Δεν πρόκειται για την μοναδική εμπορική συμφωνία την οποία υπογράφουμε αυτή τη στιγμή. Σήμερα πρέπει να πω ότι έχουμε εμπορικές συμφωνίες με όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Πριν από 8 ημέρες ολοκληρώθηκε μία νέα εμπορική συμφωνία με τη Βενεζουέλα. Ήδη έχουμε θέσει σε εφαρμογή την εμπορική συμφωνία μας με τον Καναδά. Ήδη λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για να εφαρμοστεί η εμπορική συμφωνία που έχουμε με το Περού. Ήδη εφαρμόζουμε την εμπορική συμφωνία την οποία έχουμε συνάψει με την Ελβετία και έχουμε αρχίσει συνομιλίες για μία σύμβαση ελευθέρου μπορείου και με την Τουρκία. Αυτή την εβδομάδα η υπουργό Εξωτερικών μας πήγε στην Κίνα και στην Ιαπωνία για την σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών και με τις δύο αυτές χώρες. Εγώ προσωπικά πήγα στη Ρωσία στις 22 και 23 Φεβρουαρίου για να ε, διαρρεύσω τις δυνατότητες εμπορικής συμφωνίας με την Ρωσία προσπαθώντας να συνάψουμε συμφωνία όπως αυτή την οποία θα κάνουμε και με την Τουρκία, γιατί είμαστε στην ίδια θέση την οποία βρίσκονται και οι άλλες χώρες τη Λατινική Αμερικής και της Καραβικής. Ο στόχος μας είναι να αναπτυχθούμε οικονομικά. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μελετήσει σοβαρά τις επιτυχίες που έχουμε στις χώρες της Λατινικής Αμερικής σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης και πρόοδο που επιτυγχάνουμε για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα, να εξασφαλίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, διευρύνοντας ακόμη περισσότερα την δημοκρατία. Αυτό είναι κάτι που αφορά όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, όλες τις κυβερνήσεις, όλα τα κοινοβούλια μας, τα θεσμικά όργανα και όλους τους τομείς που συνεισφέρουν στην οικονομία συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματιών και των εργαζομένων. Στα πλαίσια αυτή της προοπτικής καταβάλουμε και εμείς μεγάλες προσπάθειες για να μειώσουμε την ανεργία, την φτώχεια. Καταβάλουμε προσπάθειες για την ενίσχυση των θεσμών μας, για μία πολιτική προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, τα δικαιώματα των επιχειρηματιών κτλ. τα Και, προσφαρός, και προφανώς προσπαθούμε να έχουμε πολιτική μηδενικής ανεκτικότητας σε θέματα καταστραστήγησης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που με τις ιδιάζουσες συνθήκες που έχουμε στην Κολομβία με τις εγκληματικές οργανώσεις, με την κερίγια και με όλα τα προβλήματα που έχουμε και αντιμετωπίζοντας τέτοιου είδους εγκληματικότητα να, έχουμε τέτοια, να έχει τέτοια δέσμευση όπως έχουμε εμείς με την δημοκρατία. Και για να αντιμετωπίσουμε αυτή την ε, εγκληματικότητα, σας λέγω ότι το, η ανεκτικότητά μας για αυτούς που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μηδενική. Πρέπει να πω ότι ακόμη και δημόσιοι αξιωματούχοι ε, έχουν πάει στη φυλακή. Όταν υπάρχει θέμα δεδομένου ότι η ατιμορρησία είναι κάτι το οποίο δεν ανεχόμεθα για κανένα. Επίσης, από φέτος την 1η Ιανουαρίου ισχύει ένας νέος νόμος ε, αποζημιώσεων κατά των θυμάτων βίας. Ε, των θυμάτων συνδικαλιστικής βίας. Και έχουμε και μια πολιτική επανορθωτική, αν θέλετε, για, την, ε, για να αποδοθούν και πάλι οι γέες οι οποίες, τις οποίες είχαν στερηθεί οι, οι για χρόνια. Και με, με 25 δις δολάρια προσπαθούμε ε, φέτος να κάνουμε τέτοιου είδους πολιτική και για να μπορέσουμε να αποζημιώσουμε τα θύματα δεν ζητήσαμε τη βοήθεια κανενός. Αυτό διότι μπορέσαμε να πάρουμε πίσω από τους εξεγερμένους και τους αντάρτες και αυτούς οι οποίοι είχαν ε, με παράνομο τρόπο πάρει τις γέες ε, των γροτών μας στην Ήπεθρο, κάνουμε προσπάθειες για να αποκαταστήσουμε αυτές τις αδικίες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν απειλές, ότι υπήρξαν δολοφονίες εκ μέρους παρανόμων ε, στρατιωτικών οργανώσεων, αλλά ό,τι και να κάνουν εμείς δεν υποχωρούμε. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει και μία, θα κάνουμε και μία πολιτική επανόλθωσης ε, συλλογικά κατά όλων αυτών των συνδικαλιστών που υπήρξαν θύματα της βίας. Δεν έχουμε εμπειρία, αλλά αρχίζουμε διότι θέλουμε να αρχίσει η διαδικασία η ειρηνευτική, να επικρατήσει ειρήνη και συγνώμη μεταξύ όλων αυτών που έχουν καταστρέψει ανθρώπινες ζωές. Αυτός είναι ο στόχος μας και δεν θα αλλάξουμε. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε να γίνει ένα, έτος, κράτος ευημερία στο Περού. Και ένας από τους άξονες αυτής της ευημερία είναι η πλήρης τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πρέπει να πω με όλο το σεβασμό που σας οφείλω, ότι όλα αυτά ξεπερνούν την οποιαδήποτε υπογραφή συμφωνία. Ό,τι και να κάνουμε σε όλα τα επίπεδα, στα πλαίσια του ΟΗΕ και μπορεί να μας ελέγξουν οι πάντες, το κάνουμε θέλοντας να εξασφαλίσουμε πλήρη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οποιοςδήποτε παρατηρητής, παρόν, ευρωβουλευτής, α, Όποιο έχει έρθει στην Κολομβία τελευταία χρόνια μπόρεσαν να έρθουν σε επαφή με οποιοδήποτε εκπρόσωπο οποιοδήποτε τομέα τη κοινωνία μα. Εμεί δεν ζητούμε κανένας ε, να μα. ε, ε, να είναι συνένοχος με αυτά που κάνουμε. Θέλουμε πλήρη διαφάνεια να προχωρήσουμε. Πρέπει να πω ότι είχαμε τα τελευταία 20 χρόνια τρομερή βία στη χώρα μας. Εξαφανίστηκαν περισσότερο από ένα εκατομμύριο άτομα. Θανατώθηκαν, εξαφανίστηκαν, αλλά ο πόλεμος, ο αγώνας κατά των παράνομων ενόπλων δυνάμεων συνεχίζεται μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η δημοκρατία στη χώρα μας και να εξαφανιστούν. Γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι η αναγνώριση των, της πρόοδου που επιτέθηκε εκ μέρους του εκπροσώπου του ΔΟΕ σε θέματα νομικά, σε θέματα προστασίας των συνδικαλιστικών ε, δικαιωμάτων, διότι αυτή τη στιγμή προστατεύουμε περισσότερα από 10.000 άτομα που έχουν συνδικαλιστική ε, δραστηριότητα. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι, γι' αυτό φίλοι μας, απλώς και μόνο πρέπει να σας πω ότι εμείς σεβόμαστε τις επικρίσεις που γίνονται, σεβόμεθα αυτούς που λέγουν ότι δεν συμφωνούν με αυτή την εμπορική συμφωνία, αλλά αν τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θελήσει να το εγκρίνει, θα συνεργαστούμε μαζί του. Όχι μόνο για να υπάρχουν οικονομικά ωφέλη, αλλά για να μπορέσουμε από κοινού να κάνουμε μία πολιτική αμφίδρομο σε θέματα προστασίας των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής και την κατεύθυνση της Κολομβίας. Αλλά εάν τελικά, για κάποιο άλλο λόγο, δεν εγκριθεί αυτή η συμφωνία, επιτρέψτε να πούμε, δεν θα συμβεί και τίποτε. Το τόσο σημαντικό. Θα συνεχίσουμε να έχουμε εξαιρετικέ σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι τελικά αυτό που μας ενώνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι δημοκρατικές αξίες. Οι εμπορικές συμφωνίες είναι στρατηγικοί στον τομέα του εμπορίου. Αλλά όπως σας είπα, όλες οι συμφωνίες οι εμπορικές θα έπρεπε να έχουν ανθρώπινο πρόσωπο. Αρχίζοντας από τα παιδάκια και αρχίζοντας από την πρόσφυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστώ. Και εμεί ευχαριστούμε. Ακούσαμε λοιπόν όλους όσοι ε, συμμετέχουν ε, στο πάνελ, τους επίσημους ε, προσκεκλημένους και Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών από το Περού και την Κολομβία. Ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε με την κυρία Αλεχάνδρα Αλάισα από το Περουβιανό Δίκτυο Παγκοσμιοποίησης ε, με Ισότητα. Το έχω αυτό μεταφράσει στα αγγλικά από τα ισπανικά. Και με την κυρία Τατιάνα Ροντρίγκε από τους φίλους της γης στην Κολομβία. Η πρώτη είναι από το Περού και άλλη από την Κολομβία. Ξεκινάμε με την Αλεχάνδρα ε, για τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απευθύνω χαιρετισμό στην Αντιπρόεδρο του Περού και στον Αντιπρόεδρο της Κολομβίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους είναι εδώ. Εμείς εκ μέρους της κοινωνίας των πολιτών να παρακολουθούμε αυτή τη διαδικασία αυτή τη και θα θέλαμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για τη ε, συμφωνία αυτή. Μία πρώτη διαπίστωση και κάτι που μας ανησυχεί κατά πρώτο λόγο είναι ότι δεν είναι συμφωνίες μεταξύ ίσων. Υπάρχουν μεγάλες ασυμμετρίες μεταξύ των δύο ομάδων χωρών και θα έπρεπε η συμφωνία αυτή να χειριστεί διαφορετικά τα δύο μέρη και να επικαλεστεί ειδικέ συνθήκες ώστε να μπορέσουν ε, οι διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής να επιφυληθούν περισσότερο από αυτή την εμπορική συμφωνία. Έχω ένα παράδειγμα από τον ε, τομέα των υπηρεσιών, των χρηματοπιστωτικών ε, υπηρεσιών που είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί και διαπραγματευτεί πριν από να την αρχή της κρίσης στην Ευρώπη. Σήμερα το μοντέλο αυτό τίθεται σε αμφισβήτηση και από εσάς τους ίδιους. Εσείς υποφέρετε και δεν θα πρέπει η κρίση αυτή να πλήξει και στις χώρες των Άνδεων, το Κολομβία και το Περού που κάνουν τρομερές προσπάθειες για να προχωρήσουν, να προοδεύσουν. Δεν θα πρέπει λοιπόν να συμπεριληφθεί ένα κεφάλαιο που να μην λαμβάνει υπόψη αυτή την νέα κατάσταση και να μην λαμβάνει υπόψη τα ε, συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε εσείς μετά από την οικονομική κρίση. Νομίζω ότι αυτό είναι βασική ανησυχία δική μας και θα πρέπει ε, όσο και για την αυτό το θέμα σημαντικό για την Ευρώπη, όσο και για μας να θεωρηθεί το θέμα αυτό ώστε να μπορέσουν να μπουν και οι διάφορες διασφαλίσεις που θα μας επιτρέψουν να μην ξαναπέσουμε σε τέτοιου είδους οικονομική ε, κρίση, δεδομένου ότι δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε ούτε για εσάς ούτε για μας. Δεύτερο θέμα το οποίο μας απασχολεί και μας απασχολεί όλους εμάς και την αναφέρω. Οι οργανώσεις που παρακολουθούν αυτή τη συμφωνία θεωρούν ότι Η εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχει γίνει σεβαστή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα ε, γενικευμένων προτιμήσεων και σε θέματα εργασιακά. Θέλουμε να, να έχουμε μία συμφωνία στην οποία να υπάρχει ένα εποπτικό όργανο το οποίο να επιλύει διαφορές και να μπορεί να εγγυάται σωστούς εργασιακούς όρους για τους εργαζομένους. Επίσης, σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα, να μπορούν οι διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις να κινούν τις διαδικασίες για την προστασία των εργαζομένων οι μηχανισμοί εδώ που προβλέπονται δεν είναι αρκετά ισχυροί ώστε να, γίνονται, να, να δίδει εγγύηση στα δικαιώματα των εργαζομένων. Για θέματα εργασιακά λοιπόν, για θέματα περιβαλλοντικά θα θέλαμε να γίνουν οι σχετικές τροπολογίες ώστε να υπάρχει βελτίωση των ε, προστασίας των ε, ε, δικαιωμάτων των εργαζομένων στις ίπα ε, προβλέπονται ε, πολύ ψηλότερα τρα στάνταρ και οι κυρίως όσον αφορά τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Και αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται στην ουρά. Τελευταία, θα ήθελα να πω αυτά τα οποία είπε η κυρία Μαρισόλε Σπινόσα και να πω ότι είναι κατεπήγον η συζήτηση αυτή να γίνει στο Περού. Σήμερα είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η συζήτηση αυτή θα πρέπει να γίνει και στην ε, Βουλή του Περού, όχι μόνο για θέματα ε, που αφορούν την ε, δημοκρατία, αλλά και για θέματα τα οποία αφορούν τα εργασιακά θέματα που είναι τόσο σημαντικά για μας η κυρία Τατιάνα Ροντρίγκε ε, ε, από, τον οργανισμό Friends of the Earth, η της γης από την Κολομπία. Γεια σας σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας ε, για την οποία μας ζήτησε να κάνουμε Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2009 Παρακαλώ, αν θέλετε να σας καταλάβουν και όσοι δεν μιλούν ισπανικά, να μιλάτε πιο αργά, λέει ο πρόεδρος, για να προλαβαίνουν και οι δύστιχοι διερμηνείς. Λοιπόν, η αξιολόγηση επιπτώσεων για την βιωσιμότητα του εμπορίου που μου παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι εάν δεν υπάρχουν ε, οι κατάλληλες αλλαγές δεν θα μπορέσει να βελτιωθούν οι συνθήκες για τους εργαζομένους και για την γεωργία. Το θέμα επίσης ε, της ε, εκμετάλλευσης των φυσικών μας πόρων στο Περού και στην Κολομβία είναι πολύ σημαντικό και αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μην ε, υπάρχει εξάντληξη αυτών των πόρων με το εμπόριο το εντατικό που προβλέπεται. Γίνεται κυρίως όσον αφορά την εξορρυκτική βιομηχανία στις ε, χώρες μας, δεδομένου ότι είμαστε στην περιοχή μας χώρες που είμαστε οι πιο πλούσιες σε θέματα βιοπικιλότητας, αν θέλετε, όσον αφορά την εξορρυκτική μας δυνατότητα. Επίσης, το θέμα της πρόσβασης στο νερό. Εκ μέρους των βιομηχανιών, ε, για λόγους μόλυνσης. Είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Καθημερινά προσπαθούμε να καταπολετήσουμε το θέμα αυτό της μόλυνσης των υδάτων από τις δραστηριότητες κυρίως της εξωτερικής, εξορυκτικής βιομηχανίας. Επίσης, το θέμα των απαλωτριώσεων των γεών είναι κάτι που μας απασχολεί στην Κολομβία. Σήμερα το 40% όλης της, ε, ε, όλο του εδάφους μας ε, αφιερώνεται στην εξορρεκτική βιομηχανία. Και υπάρχουν μεγάλα προβλήματα με τα άτομα τα οποία Όπως είπε και ο εκπρόσωπος της ε, Κολομβίας, με το θέμα της αποκατάστασης ε, του θέματος ε, της απαλατρίωσης των γεών. Μία μόνον εταιρεία όμως, μία πολυεθνική από την Νότιο Αφρική έχει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των γεών που έχουν απαλατριωθεί. Επίσης, το θέμα της ε, παράνομης ε, ε, υλοτομίας, η αποψήλωση των δασών, τα κλιματικά προβλήματα. Είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν και κάνουν την τη φύση μας πιο ευάλωτη. Το περιβάλλον μας όλο και περισσότερο, το κλίμα και το περιβάλλον όλο και περισσότερο πλήττονται από διάφορες ε, βιομηχανικές δραστηριότητες, κυρίως τη μονοκαλλιέργεια, την εξορρεκτική βιομηχανία και η, φυσική η φυσική μας πόλη όρο και περισσότερο μειώνονται. Γι' αυτό οι διάφορες επενδύσεις που δίδονται στα γιγαντιαία project των πολυεθνικών είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει καθόλου την κοινωνική ανάπτυξη της κοινωνιών μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να συνεισφέρει ακόμη περισσότερο στις κοινωνικές διαμάχες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας. Τώρα λοιπόν θα ακούσουμε και την πλευρά του Κοινοβουλίου. Πάρα πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο. Πρώτος, ε, λοιπόν, πρώτα θα δώσω το λόγο στην ε, ομάδα που καταθέτει έκθεση από αυτή την Επιτροπή. Αποτελείται από τον εισηγητή και τους και εισηγητές. Και μετά θα περάσω σε άλλα όργανα του Κοινοβουλίου που παρίστανται, δηλαδή στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, στην Αντιπροσωπεία που ασχολείται με την κοινωνία των πολιτών και θα δώσω και σε άλλου το λόγο. Είναι πάρα Ε, και πρέπει κάπω να περιορίσω τον αριθμό των ομιλητών. Α ξεκινήσουμε λοιπόν κάθε ομιλητή για τρία λεπτά. Ο εισηγητή είναι ο Μάριο Νταβίδ από το ΕΛΚ και του δίνω το λόγο. Και ζητώ από τους εμπειρογνώμονες μας ε, και τους ομιλητές ε, να λάβουν υπόψη τους τις ερωτήσεις και στο τέλος θα απαντήσουν. Μάριο, έχετε το Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ το πρόγραμμα ανέφερε ότι θα γίνουν πρώτα απ' όλα, θα ληφθούν κάποια συμπεράσματα. Γι' αυτό λοιπόν ας ακούσω τα συμπεράσματα και ως συγητή σας πάρω μετά το λόγο, λέει ο κύριος Δαβίδ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε. Σε ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψή σας. Θα ήθελα να αναφερθώ ε, σε κάτι που είπε ο κύριος Γκαρτσό, ε, Αναφέρθηκε στη συνεργασία ε, για την εφαρμογή της συμφωνίας. Στις ανακοινώσεις των εμπειρογνωμόνων μου κατέστη σαφές ότι το θέμα της εφαρμογής είναι καθοριστική σημασίας. Γι' αυτό λοιπόν το δικό μου το ερώτημα είναι το εξής. Κατά πόσον σε κρίσιμα θέματα όπως είναι η ποινική δίωξη ή η διαφύλαξη ε, δικαιωμάτων ε, συλλογικών συμβάσεων. Γνωρίζουμε παρήματος χάρη ότι στην ε, Κολομβία Μόνο 4% των συναδέλφων ε, καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Και όσον αφορά στον αριθμό των επιθεωρητών ε, για την παρακολούθηση των εργατικών δικαιωμάτων και εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί. Ε, ίσως λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μία συμφωνία για να διασφαλίζεται η εφαρμογή της συμφωνίας έτσι ώστε να έχουμε την εγγύηση ότι οι δυσκολίες που αφορούν στην υλοποίηση των εργατικών δικαιωμάτων οι δυσκολίες αυτές αντιμετωπίζονται. Και κάτι άλλο, η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συμπεριληφθεί περισσότερο στην εφαρμογή. Μπορώ λοιπόν να φανταστώ και θα ήθελα να ακούσω εδώ τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων ότι πραγματικά ανεξάρτητα όργανο, όργανα συνδικάτων εργοδοτών και εργαζομένων είναι ε, έτοιμα να παρακολουθούν τις εξελίξεις ε, τόσο στην, στην Κολομβία και στο Περού όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα υπάρχει ανταλλαγή απόψεων έτσι ώστε να ε, διασφαλίζεται η διαδικασία εφαρμογής. γιατί είναι απόλυτα σαφές αν ε, στην Πολωνία, παραδείγματο χάρη, μιλήσω με έναν ε, ανθρακορίχο, ε, με έναν παραγωγό βιοκαυσίμων στην Γερμανία, με έναν ανθοπόλη στην Ολλανδία, όλοι ξέρουν περί τίνο πρόκειται. Και ίσω το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και στην Κολομβία και στο Βέλγιο να ξέρουν και αυτοί το τι ακριβώ ισχύει. Ευχαριστώ πολύ. Τρία λεπτά ακριβώ, πολύ ωραία. Περνούμε ε, Στι άλλε ομάδες. Κάθεν Μπιερδά από τους ε, Φιλόφους Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους ε, σημερινού ομιλητές. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η συζήτηση μέχρι τώρα. Θα ήθελα εγώ να εστιαστώ σε ορισμένα σημεία. Τα διασφάλιση των δικαιωμάτων, των περιουσιακών δικαιωμάτων, από ό,τι καταλαβαίνω στην Κολομβία, στην Κολομβία ε, καταγράφεται καλύτερα στο νόμο, στο δίκαιο, αλλά αυτή η δικασία παίρνει πολύ χρόνο. Εμένα με ανησυχεί το γεγονό ότι οι εξαιρετικέ εταιρείε είναι έτοιμε με το που ε, η συμφωνία. Θα κινηθούν πιο γρήγορα από όσους ε, ε, λάβουν αυτή την αποζημίωση ή πάρουν τη γη τους πίσω. Ακούσαμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι οι αυτόχθονες, ε, υπάρχουν αυτές οι ανισορροπίες μεταξύ ας πούμε, των αυτοχθόνων ή της, ε, της φύσης του φυσικού περιβάλλοντος και των οικονομικών φορέων. Μιλήσατε για το δίκαιο εμπόριο και εγώ θα ήθελα να ακούσω κύριε Επίτροπε πώς το, πώς το υλοποιούμε αυτό και πώς θα συνδράμουμε την Κολομβία και το Περού για να προστατεύσουμε τις να τις προστατεύσουμε από τις ε, εταιρείε ή να προστατεύσουμε τις εταιρείε μας από επικίνδυνες καταστάσεις. Μετά, η προστασία από τη μόλυνση του περιβάλλοντος είναι σαφώς ε, ε, ζητήματα που μας προβληματίζουν. Και εγώ θα ήθελα να δούμε αυτό το say what you pay, αυτή τη γνωστή ρίση και στις δικές μας επιχειρήσεις για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς πληρώνουν οι επιχειρήσεις μας. Και δεν πάμε απλώς ε, να εξορίξουμε και φέρνουμε πίσω τις ε, πρώτες ύλες. Πρέπει να ε, ενθαρρύνουμε και να βοηθούμε τις επιχειρήσεις επιτόπους, εκείνη τη χώρα δηλαδή, να ε, επεξεργαστούν για τις πρώτες ύλε και να παραδώσουν το τελικό προϊόν. Αυτό θα τους βοηθήσει γενικότερα. Με προβληματίζει ακόμα αυτή η συμφωνία. Θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ από τους ε, συντηρητικούς Γιάννη Τζαράντιου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Ντεγιούχτ για τις ε, πολύ τολμηρές και ξεκάθαρες ε, απόψεις του, καθώς και τους αντιπροέδρους για τις παρουσιάσεις τους. Λαμβάνοντα υπόψη όλους τους προβληματισμούς και τις αμφιβολίες, ε, πρέπει να πω ότι εγώ και η ομάδα μου θεωρούμε αυτή τη συμφωνία μια ευκαιρία, μια θετική εξέλιξη. Και θέλουμε να τονίσουμε ότι αυτή η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μπορεί να ανοίξει το δρόμο και για την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κάτι που για μας είναι πολύ σημαντικό. Θεωρούμε ότι θα ε, ευνοήσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε όλες τις πλευρές και αυτό πολύ θετικό και τελικά θα οδηγήσει σε σύγκληση στα εργασιακά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά πρότυπα. Με απλά λόγια, Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα μέσο για την προώθηση της σταθερότητας, της ευημερίας και συνεργασίας σε άλλους τομείς που συνδέονται με το εμπόριο, όπως η έρευνα και ανάπτυξη, η καινοτομία, ο εξεχρονισμός και παρόμοιοι τομείς. Γι' αυτό το λόγο, σε γενικές γραμμές, στηρίζουμε ιδιαίτερως ε, αυτή τη συμφωνία. Τώρα, για τα λοιπά, πρέπει να πω ότι κατανοώ την κατάσταση. Ε, εδώ μιλάμε για δημοκρατικές χώρες, δημοκρατικές κοινωνίες, χώρες που έχουν ε, περάσει δύσκολες ε, περιόδους στο παρελθόν, αλλά τώρα έχουν εκλεξ, ε, ε, δημοκρατικά εκλεγμένους ε, αρχηγούς που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις προκλήσεις και να κάνουν ό,τι μπορούν για να ευνοήσουν ε, τις συνθήκες στις χώρες τους. Και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να βλέπουμε τους εταίρους μας στην Κολομβία και το Περού ως ισότιμους εταίρους και κυρίαρχα κράτη. Αυτή είναι η καλύτερη προσέγγιση αυτή τη στιγμή. Αυτά είχα να πω προς το παρόν. Ούτε καν ε, υπερεύει το χρόνο μου. Συνοψίζοντας μπορώ να πω ότι εγώ και η ομάδα μου ε, διακύμεθα θετικά. Ευχαριστούμε σκιώδης συζητητή ε, των Πρασίνων. Σωσέφ δεν είναι εδώ. Αλεξάνδρο θα τον αντικαταστήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Πολλά έχουν ήδη υποθεί για τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Δεν θέλω να επανέλθω λοιπόν, ακόμα και αν είναι ιδιαίτερο σημαντικό ω ε, ζήτημα. Βεβαίω ε, και ε, προσβλέπω σε ε, ενεργό συμμετοχή σα και δέσμευσή σας να διασφαλίσετε ότι τα μέτρα αυτά θα... και τα δικαιώματα όλα αυτά θα γίνονται σεβαστά. Δυστυχώς η ιστορία δεν δίνει πολύ αξιοπιστία στην Επιτροπή σε αυτό το επίπεδο γιατί τη στιγμή όπου υπήρξαν οι περισσότερες δολοφονίες στην Κολομβία η Επιτροπή είχε αρνηθεί όχι να, να ανακαλέσει την ε, συμφωνία, αλλά να κάνει μια έρευνα, να διερευνήσει αν ε, θα μπορούσε να υπάρξει ανάκληση ενδεχομένω τη απόφαση. Δεν ξέρω λοιπόν τι θα μπορούσε να διασφαλίσει ότι στο μέλλον η Επιτροπή θα είναι πιο αξιόπιστη από ό,τι στο παρελθόν. Τώρα για τη συμφωνία Έχω ορισμένα ερωτήματα για, τις, για τους εκπροσώπους της Κολομβίας και του Περού. Πρώτον, πώς ε, ε, βλέπετε το γεγονός ότι η Ευρώπη μπορεί να εξάγει ε, γάλα, για παράδειγμα, με, με ποσόστοση που θέτει αναμφιβόλο βεβαίως πολλές μικρές επιχειρήσεις στην χώρα σας. Ήταν δύσκολο στοιχείο των διαπραγματεύσεων. Πώ λοιπόν θα διαχειριστείτε στην χώρα σας σε τέτοιε διατάξεις. Τώρα για τι υπηρεσίες. Έχουμε την φιλελευθερωποίηση των υπηρεσιών στη χώρα σας, ιδιαίτερα ισχυρή σε ό,τι αφορά ε, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, νερό. Ξέρουμε δυστυχώ, η εμπειρία μα δείχνει ότι ορισμένοι μεγάλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι δεν διασφαλίζουν το γενικό συμφέρον εφόσον έχουν αποκτήσει τις υπηρεσίες που θέλουν. Τι ακριβώς λοιπόν έχετε στα χέρια σας για να, ε, ως εχέγγυο. Τέλος, για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και υπηρεσίες ε, ετέθη ξεκάθαρα. Ε, το ερώτημα το απευθύνω προς εσάς κύριε Επιτροπέ. Τι ακριβώς θα κάνετε και γενικά η Επιτροπή, η Ευρώπη για να για να προστευθεί από ενδεχόμενα επικίνδυνα απόβλητα που προέρχονται από τέτοιες χώρες με τις οποίες έχετε ε, συνάψει συμφωνίες. Ε, εδώ και τα τελευταία χρόνια ε, θέλαν να υπάρχουν συμφωνίες για να αποφύγουν αυτά τα τοξικά προϊόντα εντό εισαγωγικών. Ευχαριστώ. Um, on Τώρα, Εκ μέρου Ευρωπαϊκή ε, Ενωμένη Αριστερά, ο κύριος Χέλμουντ Σόλτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και ε, τους Αντιπροέδρους ε, και όλους τους άλλους που μας έδωσαν τη δυνατότητα να κατανοήσουμε ένα περίπλοκο θέμα. Επίσης χαίρομαι για το ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον εδώ στην Έτσο και αυτό δείχνει ότι η γνώση πολλών εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, των ε, συνδικάτων. Η γνώση λοιπόν αποδεικνύει ότι αυτοί έχουν όλοι ασχοληθεί με τη μακρά ιστορία του όλου κινήματος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει λοιπόν να εξετάσει ε, το πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι νέες ε, στρατηγικές των κυβερνήσεων και στο Περού και στην Κολομβία είναι στρατηγικές για την αντιμετώπιση του παρελθόντος. Γι' αυτό λοιπόν καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι διαφανής στην προσέγγιση της. Και ως εκ τούτου πρέπει να ερωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τι πραγματικά μπορεί να γίνει. Να γνωρίζουμε λοιπόν ότι ε, ποιες είναι οι πραγματικές ανησυχίες της κοινωνίας των πολιτών. Οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, ε, τα εργατικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των δημοσιογράφων, αυτά είναι πολύ σημαντικά για να μπορεί κανείς ε, να τα αντιμετωπίσει και να πρέπει να τα αντιμετωπίσει στη χώρα του. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να τεθεί. Ε, υπάρχει λοιπόν και κάτι που είναι σωστό, ότι διαπραγματευόμαστε σε επίσης όρις. Ε, τους αντιμετωπίζουμε ε, ως ίση προσίσων. Κατόπιν τούτου, ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα κάτω από αυτό το πρίσμα. Και τέθη ήδη το ερώτημα ποιες, τι, δυνατότητες, δυνατότητες έχει ας πούμε ένας ε, Έλληνας ε, συνδικαλιστής ε, και επιχειρηματίας μικρομεσαίος στην κρίση την οποία βιώνει να έρθει σε επαφή με το Περού για να ενημερωθεί πώς μπορεί να επιβιώσει. Αυτή λοιπόν η συμφωνία πώς μπορεί να προσαρμοστεί στην οικονομική πραγματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Περού και στην Κολομβία. Ε, πώς μπορούμε να μεταφέρουμε αυτή την εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ήδη αναφέρθηκε ο Αντρακορίχος στην Πολωνία, αλλά πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα στις ανατολικές χώρες, στην Ελλάδα ε, και σε άλλες χώρες και όχι μόνο να αναφερόμαστε σε μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις και κάτι άλλο ακόμα. Ξέρω βέβαια ότι περνάει ο χρόνος ασχολούμεθα με το θέμα αυτό σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να ακούσουμε πιο προσεκτικά τα δικαιώματα των αυτοχθόνων, τα δικαιώματα των πέννητων στη χώρα. Και θέλω να πω το εξής, η άποψη, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχει ε, λάβει οριστική μορφή όσον αφορά αυτή την Συμφωνία Ελεύθερων Εμπορικών Ανταλλαγών. Πρόεδρος, πριν δώσω το λόγο και σε άλλα μέλη της Επιτροπής, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Σαλαφράγκα από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και μία ερώτηση στον Επίτροπο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε ποια είναι τα πλαίσια μέσα στην οποία εγγράφεται αυτή η εμπορική συμφωνία. Πρώτη συμφωνία, πρώτη γενιά που συνάψαμε, αυτό το οποίο τόνισε είναι η συνεργασία και αναπτυξιακή βοήθεια. Τη δεύτερη, τεχνολογική και επιστημονική σύνδρομη. Τρίτη, η ρήτρα εκδημοκρατισμού και η οικονομική βοήθεια. Και αυτή η τέταρτη συμφωνία, τέταρτης γενιάς, ε, προοδευτική απελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών. Εγώ ήμουνα, ε, συμμετείχα στις δύο ε, εμπορικές συμφωνίες που είχαμε με άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής και πρέπει να πω ότι πραγματικά ε, συνεισέφεραν στη βελτίωση του ΑΕΠ όπως είπε και ο Επίτροπος για την Περού και την Βολιβία. Ο στόχο είναι διπλός. Οι δύο χώρες αυτές να παίξουν στην ε, ε πρώτη εθνική, αν θέλετε, στην κατηγορία κρατών πρώτης εθνικής όσον αφορά τι εργασίες με τρίτες χώρες, δεδομένου ότι πρόκειται για συμφωνίε μεταξύ ίσων μερών. Δηλαδή, πρόκειται για συμφωνίες οι οποίες προβλέπουν η ισοδυναμία μεταξύ των δύο μερών παρά το γεγονός ότι λαμβάνονται υπόψη σωστά οι ασυμμετρίες όπως λέγονται. Δεδομένου ότι η απελευθέρωση των βιομηχανικών προϊόντων ε, ένθεν και ένθεν γίνεται για 100% των προϊόντων με διάφορες ε, ρήτρες και η δημοκρατική ρήτρα είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στην περίπτωση του Περού του Φούτζι Μόρι είχαμε μία λιγότερο ε, χτενισμένη στις λεπτομέρειες συμφωνία αν θέλατε και σήμερα δεν θα μπορέσαμε να την κάνουμε. Δεν θα πρέπει να πούμε εμείς στους ε, φίλους μας των κρατών της Λατινικής Αμερικής δεν θα πρέπει να έχουμε αυτή την υπεροψία να τους πούμε εμείς τι είναι καλύτερο για αυτούς και τι δεν είναι. Είναι δημοκρατικές χώρες, έχουν εκλεγμένα όργανα, ας ακούσουμε τι έχουν να μας πούνε, αλλά θα πρέπει οι εκπρόσωποι των ε, πολιτών των κρατών αυτών να μας πούν τι τους αρέσει ή όχι και τι, με τι συμφωνούν ή όχι. Κύριε Πρόεδρε, δεν πιστεύετε ότι χάνουμε την αξιοπιστία μας όταν έχουν περάσει δέκα χρόνια, ε, δύο χρόνια μετά από τις συμφωνίες της Μανδρίτης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιμένει τόσο καιρό για να πει ποια είναι η άποψή του για τις συμφωνίες αυτές που έχουμε συνάψει εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ε, χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ευχαριστώ πολύ. Ξέχασα να σας πω ότι ο κύριος Ελαφράκη προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Περνάμε στους επόμενου ομιλητέ Richard Χάρτ από τους Σοσιαλιστές. Δεν ανήκει στην Επιτροπή, αλλά καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. και θα ήθελα να πω στον Αντιπρόεδρο Καθόν, ε, ε, λατρεύουμε τη χώρα σας και το λαό της. Και βεβαίως και εμείς επιθυμούμε την ε, ειρήνη στη χώρα σας. Τώρα, υπήρξαν τρεις δολοφονίες συνδικαλιστών τον Ιανουάριο μετά από πυροβολισμούς και βεβαίως ε, και ε, βασανιστήρια στα στην νύχτα της 9ης ε, Ιανουαρίου καθώς ε, πήγαινε προς τη δουλειά του άνθρωπος και έτσι έχουμε φτάσει σε έναν ε, υπερβολ... τεράστιο αριθμό, τρομακτικά τεράστιο αριθμό. Τι νομίζετε ότι μπορεί να γίνει για να αναστραφεί αυτή η περίπτωση. Είπατε ότι ότι θα παρακολουθήσετε την παράνομη κατασκοπία από την ε, ε, κολομβιακή κυβέρνηση και αυτό δημιούργησε αμφιβολίες για το κατά πόσο η Κολομβία μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο ε, εταίρο σε αυτή τη συμφωνία. Τι βρήκατε με βάση την έρευνά σας ο εκπρόσωπος των Μένων Εθνών στην Υποκοτά είπε ότι συνεχίζεται η παράνομη κατασκοπία. Συμφωνείτε με τον Αντιπρόεδρο Γαθών, σε αντίθεση με τα όσα είπατε εσείς, είπατε ότι ε, φεύγουμε από την, ε, απομακρυνόμαστε από την Κολομβία. Αν η συμφωνία αυτή ε, παραταθεί, θα, είμαστε, θα εξακολουθήσουμε να είμαστε καλοί φίλοι με την Κολομβία. Προ τον ΔΟΕ, σα ευχαριστώ, αλλά πραγματικά υπάρχει μεγάλη διαφορά με αυτά που λέει και η κυβέρνηση για τα συνδικά συνδικάτα και γι' αυτό που λένε τα ίδια τα συνδικάτα. Και τόσο αναφέρονται για την σύμβαση του ILO 97 και 87. Αποδέχεστε ότι είτε πάρουμε τα στοιχεία της κυβέρνησης, είτε των σωματείων, είτε έχουμε 93%, είτε 98% ατιμορρησία σε ό,τι αφορά τους συνδικαλιστές. Και κύριε Καρθόν, Βεβαίως και θέλουμε αυτά που προσφέρετε, αλλά κατανοείτε ότι όταν μιλάμε για δολοφονίες ε, ε, συνδικαλιστών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, θα αυξηθεί και η πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν υπάρχουν καταδίκες για αυτούς τους φόνους. Και κατανοείται ότι στο ποινικό δίκαιο, ή το δίκαιο των ε, θυμάτων, όταν επιστρέφουν όλοι αυτοί στις χώρες τους, ή αν δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να επιστρέψουν στις χώρες τους και στα εδάφη τους, αυτό θα ε, δώσει καλύτερη εντύπωση στην Ευρώπη ε, για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα αποδέχεστε όλα αυτά. <clears throat> Ο κύριος Γιούργεν Κλούτε από την Επιτροπή ε, Νοτικής Αριστεράς, που και αυτός βέβαια δεν είναι μέλος της Επιτροπής μας, παρόλα αυτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να υπογραμμίσω αυτά που μόλις τώρα είπε ο συνάδελφος από την ομάδα των Πρασίνων. Δεν θέλω να το επαναλάβω, αλλά ε, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου καθεστώτος ε, υπήρξαν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μπορούσε να ε, ανασταλεί αυτό το καθεστώς. Κάτι τέτοιο όμως ε, δεν συνέβη. Και αυτό δημιουργεί μεγάλη αμφιβολία για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα γίνει στο μέλλον. Δηλαδή αυτό το καθεστώς, ε, κύριε Ντεγκούτ, πώς θέλετε να το ξεκαθαρίσετε ότι αν τελικά συνεχιστεί αυτή η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πώς θα αντιδράσετε, ε, πώς θα προσπαθήσετε να είστε αξιόπιστος απέναντι στην κοινωνία των πολιτών και κάτι άλλο. Ο κύριος Λασάν το είπε, δηλαδή πράγματι υπάρχει το φαινόμενο ε, γεών που απαλωτριώθηκαν και θα επιστραφούν. Σωστό αυτό. Οι συζητήσεις που είχα με εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών και με συνδικαλιστές με οδήγησαν στο να καταλήξω στο εξή ότι επιστράφηκε, επιστράφησαν γέες που ανήκαν στην κυβέρνηση, όχι αυτές που είχαν υφαρπαγή Μιλάμε για 60.000 οικόπεδα που πρέπει να επιστραφούν. Μέχρι τώρα όμως έχουν επιστραφεί μόνο 11.000 από την κυβέρνηση Σάντος. Και γι' αυτό λοιπόν ε, τίθεται το ερώτημα, τελικά πώς θα τα κατορθώσετε, πώς θα κατορθώσετε να φτάσετε τις 60.000 από τις 11. Και μία τελευταία παρατήρηση. Στην Κολομβία το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο άρχισε, και καλό αυτό, το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. Άρχισε λοιπόν το δικαστήριο να επεξεργάζεται υποθέσεις σε ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό όμως μας ανησυχεί. Ο πρόεδρος Κολομβίας, Σάντος, επέκρινε δρυμύτατα για το θέμα αυτό το ανώτο συνταγματικό δικαστήριο και τίθεται το εξή ερώτημα. Αυτό τώρα τι συνέπειες θα έχει. Δηλαδή τι γίνεται. Έχουμε τον αρχηγό της κυβέρνησης ο οποίος επικρίνει, δρυμύτατα μάλιστα, αυτή την όχι μόνο ορθή, ορθότατη δουλειά του ανώτατου συνταγματικού δικαστηρίου. Τι έχετε να πείτε από αυτού. Και τέλος, ο κύριος Μάια, επίσης από την ΚΟΕ, που και αυτός ε, δεν είναι εδώ μέλος της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε Γαρθών, σας Είπα και προσωπικά όταν επισκεφθήκαμε τις χώρες των Άντων και εσάς και τον πρόεδρο Σάντος, ποια είναι η θέση της κοινοβουλευτική μου ομάδα σε σχέση με αυτή τη συμφωνία. Σα είπα ότι η συμφωνία αυτή είναι αρνητική, όπω σα το είπαμε και τότε. Για δύο λόγου. Πρώτα απ' όλα, και συμφωνώ με τις παρεμβαίνουσες από την ε, κοινωνία των πολιτών, διότι δεν λαμβάνουν υπόψη τις ασυμμετρίες. Σύμφωνα με το PNUD, Μόνο η Αγγόλα και η Αϊτή έχουν περισσότερες ανισορροπίες και προβλήματα από τη δική σας χώρα. Πράγμα που σημαίνει ότι η παρουσία των πολυεθνικών, των καναδικών, των βορειοαμερικανικών και των ευρωπαϊκών ε, εταιριών ε, όλο και περισσότερο ε, γίνονται ιδιοκτήτριες γης και κλέβουν πλούτο από τις χώρες σας. Από οικονομικής λοιπόν πλευράς και όσον αφορά τα δικαιώματα των, ε, του λαού της Κολομβίας είναι αρνητική αυτή η συμφωνία και θα αυξηθούν οι ασυμμετρίες και τα προβλήματα αντί να μειωθούν. Εάν δεν λαμβάνουν, δεν ληφθούν υπόψη αυτά τα θέματα, όλο και περισσότερες ανισότητε και φτώχεια θα έχουμε. Στην περίπτωση της Κολομβίας, κύριε Αντιπρόεδρε, είχαμε την δυνατότητα να σας πούμε στη συνάντηση που είχαμε με τους εκπροσώπου της κοινωνίας των πολιτών εκεί, ότι ο απολογισμός σε σχέση με το τι γίνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ακόμη αρνητικό. Αρνητικό όσον αφορά την ασφάλεια των πολιτών την ασφάλεια των αυτοχθόνων, των γυναικών και των συνδικαλιστικών εκπροσώπων. Κατά άποψή μα, λοιπόν, υπό αυτέ τι συνθήκε δεν θα πρέπει να υπογραφεί εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η συμφωνία. Ελέγχθη επίση εδώ ότι θα πρέπει να αφήσουμε τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα, να αποφασίσουν. Α ε, ενημερωθούν, να συμμετάσχουν συνεδριάσει και μετά α θέσουν τι ε, συμφωνίε σε δημοψήφισμα για να δούμε ποια είναι η άποψη των πολιτών. Εάν όμως περιοριστούμε μόνο στην ενέργεια της κυβέρνησης χωρίς διαβούλευση και χωρίς διαφάνεια, δυστυχώς δεν μιλούμε για απόφαση του ε, λαού του Κολομβίας του Περού, αλλά των κυβερνώντων τους. Πιστεύω λοιπόν ότι εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το πιο σωστό είναι, θα ήταν να απορρίψει την επικύρωση αυτών των συμβουλίων όπως θα πρέπει να κάνουν και 27 βουλές μας. Πίτερ Πίτερ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Μια παρατήρηση, γιατί βλέπω ότι έχουν πει πολλά οι συνάδελφοι από την αριστερή πτέρυγα και εγώ ε, νιώθω την υποχρέωση να εκφράσω την ε, αμέριστη στήριξή μου προς αυτή τη συμφωνία. Είμαι πεπισμένη στην προκειθετική εξέλιξη. Θέλω να συγχαρώ τις κυβερνήσεις της Κολομβίας και του Περού για την πρόοδο που έχουν σημειώσει την τελευταία δεκαετία και κυρίως και κυρίως τα τελευταία χρόνια οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση και είμαι πεπισμένος ότι αυτή η συμφωνία θα τις βοηθήσει να επιταχύνουν ε, αυτή, τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, ε, την οικονομική ανάπτυξη και την ε, μεταχείριση των Ιθαγενών. Βεβαίως πρέπει να κοιτάξουμε και την άλλη πτυχή της εξίσωσης. Θέλω εγώ θα στηρίξω ε, αυτή τη συμφωνία για αυτόν τον λόγο. Ευχαριστώ. Μην ε, παραπονιέστε. συνήθω ε, η αντιπολίτευση είναι πιο ισχυρή στη δράση τη από ότι η πτέρυγα που συμφωνεί. Α περάσουμε τώρα στι απαντήσει. Θα τα πάρω με τη σειρά. Άντριαν Φαντινχόβεν από την Business Europe. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε στις ε, ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να απαντήσω στον κύριο Χάλιτ. Να σας πω ότι στη δική μου την ομιλία εγώ δεν είπα ότι κατά την άποψή μου η Κολομβία και το Περού και όλα τα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σέβονται πλήρω ε, τις προδιαγραφές του διεθνού Γραφείου εργασία. Η Κολομβία, το Περού και τα 27 κράτη-μέλη πρέπει όμως ε, να σέβονται τις ε, δεσμεύσει αυτέ του Γραφείου εργασία. γιατί εμεί πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές οι διεθνεί συμβάσεις είτε στον τομέα τη εργασία, είτε στον τομέα του περιβάλλοντος, είτε στον εμπορικό τομέα. Το δεύτερο θέμα που υπογράμμισα είναι το εξή. Κατά την άποψή μου, αν τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει να λάβει μέτρα απέναντι στην Κολομβία ή απέναντι στο Περού ή αντίθετα η Κολομβία ή το Περού απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά οποιοδήποτε κεφάλαιο της συμφωνίας είτε το εμπορικό είτε τα θέματα που έχουν σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη εμείς προτείνουμε όποιος πάρει αυτή την πρωτοβουλία να έρθει σε επαφή με τους κοινωνικούς εταίρους. Να μπορούν οι κοινωνικοί εταίροι να ε, εκφράσουν την άποψή τους ε, κατά πόσον ε, είναι συμβατές αυτές οι πράξεις είτε με τα εμπορικά κριτήρια είτε με τα κριτήρια περί βιώσιμης ανάπτυξης. Ο Εδουαρδό Εστέβες, πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχει καλή θέληση και καλές προθέσεις. Και εκ μέρους θεσμικών οργάνων ή ατόμων όπως ο κύριος Γαρσόν που θεωρώ φίλο. Δυστυχώς όμως πρέπει να βασιστούμε σε γεγονότα και αριθμούς. Είπαμε, αναγνωρίζουμε ότι έχει υπάρξει κάποια πρόοδος. Αλλά είναι ανεπαρκής, να είμαστε σαφείς. Επίσης, είχαμε την δυνατότητα να ζητήσουμε την άποψη των εργαζομένων στο Περού σε μια παρεμφερή υπόθεση. Κυρίως μας απασχολούν ε, θέματα τα οποία νομίζω ότι δεν λαμβάνονται υπόψη στην συμφωνία που συζητούμε. Ένα παράδειγμα. Η αύξηση του ΑΕΠ για μας δεν είναι εγγύηση ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση για αυτή. Ευτυχώς στη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια έχουμε αύξηση του ΑΕΠ ακόμη και μεγαλύτερη από αυτή τον ΗΠΑ, του Καναδά και πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ωφελεί αλλού τους πολίτες. Υπάρχει ένα θέμα αδικίας από το οποίο υποφέρουν όχι μόνο οι πολίτες των δικών μας χωρών, αλλά όλοι οι πολίτες της Λατινικής Αμερικής. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι οι πολιτικές που αναπτύσσονται και αυτή η εμπορική συμφωνία θα τροφοδοτήσει αυτή την κατάσταση, δεν θα βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και ζωής των εργαζομένων πέραν της ε, βούλησης των δύο κυβερνήσεων. Καλή βούληση έχουν, αλλά τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Ράσιο Γκίδο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω σε τρεις ε, ομιλητές που αναφέρθηκαν στον ΔΟΕ. Ένας από τους πρώτους αναφέρθηκε στο τι είδου έλεγχος μπορεί να γίνει για τα θέματα τα εργασιακά βασικά της ε, συμφωνίες τις εργασιακές. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα στην παρέμβασή μου σύντομα για την δυνατότητα να αναφερθεί κανεί στις εκθέσεις των εποπτικών οργάνων του ΔΟΕ όπου γίνεται αναφορά στα συνδικαλιστικά θέματα όπως ε, ε, κυρίως το θέμα 1787, περίπτωση που παρουσιάστηκε στα εποπτικά όργανα και καθώς και τις αποφάσεις οι οποίες ε, αφορούν τέτοιου είδους θέματα διώξεως συνδικαλιστικών οργάνων. Το ίδιο όσον αφορά και τις εγγυήσεις στην εργασία. Και αναφέρομαι στις συλλογικές συμβάσεις. Στις παρατηρήσεις του Νοεμβρίου του 2011 η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σημειώνει με ικανοποίηση ότι εγκρίθηκε νόμος για να αποφευχθεί η επιβολή συμβολικών ε, συμβάσεων. και το γεγονός ότι επιβάλλονται κυρώσεις συνδικαλιστικά όργανα. Επίσης, κάτι που αναφέρθηκε και αφορά τις επιθετικές εργασία. Έγινε το Φεβρουάριο του 2011 μια αποστολή εκ μέρου του ΔΟΕ και ενημερωθήκαμε για το ότι έχουν διοριστεί πολλοί επιθεωρητέ εργασία. Κάποια άλλη ομιλήτρια αναφέρθηκε στο τι μπορεί να γίνει για να λαμβάνουμε υπόψη τα ανησυχίε ε, για τις οποίες μας μίλησαν οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Πρέπει να σας πω ότι σε εθνικό και διεθνές επίπεδο οι εργόμενοι των εργαζομένων μπορεί να μας κάνουν σχόλια όχι μόνο για την ε, συμβάσεις ή για την συνδικαλιστική ε, ελευθερία, διότι όπως είπε και αντιπρόεδρος του Περού εκ μέρους της Επιτροπής υπάρχει έκθεση η οποία διαπιστώνει με ικανοποίηση προστάθειες που γίνονται για να ληφθούν υπόψη όλες οι κοινότητες αυτόχθονων πολιτών. Πιστεύω λοιπόν ότι όχι μόνο θέματα ε, ε, ότι όλοι οι πολίτες, ακόμη και οι τεχνικοί για οποιοδήποτε θέμα, μπορούν να προσφύγουν και να ζητήσουν τη συνδρομή του ΔΟΕ. Επίσης, κάποιος ανέφερε ε, το θέμα των αριθμών που εμείς ε, παρουσιάζουμε είπε ότι υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις όσον αφορά τις δολοφονίες συνδικαλιστικών μελών καθώς και τις καταδικαστικές αποφάσεις των τελευταίων ε, ετών. Εγώ είπα ότι το 2001 είχαμε μία τέτοια καταδικαστική απόφαση, ενώ το 2010 περίπου 400 εκφράζουμε τη λύπη μας για τις πράξεις βίας κατά των συνδικαλιστικών και τις δολοφονίες που λαμβάνουν χώρα εδώ και χρόνια. Λαμβάνουμε υπόψη αυτά τα γεγονότα και έχουμε τις στατιστικές μας και πρέπει να πω ότι εκτιμούμε όλες τις, τα πρακτικά τεχνικά και νομοθετικά μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση για να μπορέσει να ε, μειώσει τον αριθμό των ε, δολοφονιών και είμαστε υπέρ όλων των μέτρων που λαμβάνονται για την καταδίκη των ενόχων. Καταδικάζουμε τη βία εκ μέρους του ΟΗΕ. Ευχαριστώ. Τώρα η Αντιπρόεδρος Μαρισόλ Εσπινόσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη προσοχή σημείωσα όλες τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι εκπρόσωποι σας εδώ. Και εγώ θα ήθελα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τονίσω ότι η κυβέρνησή μου ενεργεί, λαμβάνοντας δεσμεύσεις και ενεργεί με διαφάνεια. Θα θέλω όλα αυτά να σας πω ότι λαμβάνονται υπόψη, θέλουμε όντως να είμαστε ένα κράτη, κράτος δικαίου και λαμβάνω υπόψη για τα εργασιακά θέματα τις ανησυχίες που εξέφεραν κάποιοι ευρωβουλευτές. Όντως, συμφωνούμε και εμείς ότι σε θέματα εργασιακά θα επικυρώσουμε όλες τις ε, ε συμβάσεις που πρέπει στα πλαίσια της ΔΟΕ και πρέπει να πω ότι η κυβέρνησή μας έχει δώσει στο Υπουργείο Εργασίας μεγάλες εξουσίες. Το Υπουργείο Εργασίας παλιά ήταν μόνο παρατηρητής και απλώς θεατής όλων των εργασιακών διαφορών. Σήμερα πρέπει το Υπουργείο μας να είναι πιο ενέργο. Και εμείς θα επαγρυπνούμε ώστε να γίνονται σεβαστά τα, δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτό δεν είναι μόνο υπόσχεση που δώσαμε στην προεκλογική μας εκστρατεία. Είναι ένα αίτημα μόνιμο και λαμβάνουμε υπόψη τους ε, νόμους τους οποίους ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΔΟΕ και τους οποίους επεξεργαζόμαστε ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στην τομέα αυτό με τους εργαζομένους στο Περού. Δεδομένου ότι έχουμε εδώ τον Υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, θα ήθελα να τους δώσετε το λόγο για να μιλούσουν για τα θέματα τα χρηματοπιστωτικά. Καθώς και το θέμα του ύδατος που απασχόλησε τις εκπροσώπους της ε, ε, κοινωνίας των πολιτών. Εδώ όμως δεν έχουμε να κάνουμε με τα θέματα τα οποία αφορούν την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση και άλλα τέτοιου τους θέματα. Έχουμε να κάνουμε μια εμπορική ε, συμφωνία, αλλά πρέπει να πω ότι η κυβέρνησή μου είναι εγγυήτρια των προάσπισης των μικρών δικαιωμάτων. Εδώ θέλω να σας ε, πω κάτι γιατί η σοκολάτα. Η σοκολάτα Πιέρ Μαρκολίνη που την ξέρετε εδώ στο Βέλγιο γίνεται με κακάο κρυόλιο από την περιοχή μας, από την περιοχή Πιούρα στο Περού και από μικρούς παραγωγούς και είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών μικρών παραγωγών μας που πέρασαν τα σύνορα και φτάσαμε εδώ στο Βέλγιο. Μαζί λοιπόν ενωμένοι από την τσοκολάτα Μαρκολίνη εξαντλήσετε το χρόνο που σας είχε δοθεί. Ε, θα μπορούσα να δώσω το χρόνο που υπολείπεται ε, στα υπόλοιπα μέλη της ε, αντιπροσωπείας του Περού. Δύο λεπτά σε κάθε ένα από εσάς. Παρακαλώ. Ο κύριος Δεσίλβα, γεια σας. Ευχαριστώ πρόεδρε που μου δίνετε χρόνο. Για το Περού αυτή η εμπορική συμφωνία είναι μια ευκαιρία, ευκαιρία για τους πιο φτωχούς. Και όπως μόλις τώρα είπε η Αντιπρόεδρος, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τα προϊόντα τους, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλήσαμε για το κακάο, και να τα εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε πόσο οι εξαγωγές έγιναν η κινητήρια δύναμη της οικονομίας μας. Πέρσι είχαμε αύξηση του 32% των εξαγωγών μας. Προστιθέμενη αξία μεγάλα και χιλιάδες Περουβιανοί που δεν είχαν τη δυνατότητα να δουλέψουν στο παρελθόν σήμερα ε, δουλεύουν στην εξαγωγική αλυσίδα των προϊόντων μας. Η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τις ε, εξελίξεις αυτές ώστε η φτωχή, όπως όχι οι φτωχοί Ευρωπαίοι, γιατί οι φτωχοί ε, Ευρωπαίοι για μας είναι η μέση τάξη στο Περού. Μιλάμε για τους φτωχούς φτωχούς, τους πραγματικούς που δεν έχουν πρόσβαση σε ε, αξιοπρεπή δουλειά. Αναφέρθηκε το θέμα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και στο θεωρούσε ότι τοξικά προϊόντα ευρωπαϊκά φτάνουν στο Περού. Εμείς είμαστε ήρεμοι διότι έχουμε ένα από τα πιο ασφαλή και σταθερά τραπεζικά συστήματα του κόσμου. Όταν ε, άρχισε η κρίση στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ κανένα πιστοτικό ίδρυμα δεν επηρεάστηκε στο Περού, δεδομένου ότι υπάρχει αυστηρός έλεγχος του τι ακριβώς γίνεται στον τραπεζικό τομέα. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στην δυνατότητα η εμπορική αυτή συμφωνία να περάσει από το Κογκρέσο, τη Βουλή μας. Στο σύνολο θα περάσει η συμφωνία από το Κοινοβούλιο και Πρέπει να πω ότι υπάρχουν εκπρόσωποι όλων των ε, κοινοτήτων και των ε, αυτόχθανων κοινοτήτων της χώρας μας που εκπροσωπούνται στη Βουλή μας που ζητάει αυτό το θέμα. Ο Υπουργό Περιβάλλοντος Πουλγκάρ Βιντιλβάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό μόνο για να ανταποκριθώ ε, στις ανησυχίες που εκφράστηκαν για τα στάνταρ που αφορούν το κλίμα. Όπως είπε και ο κύριος ε, Σαλαφράγκα θα πρέπει να δούμε στο σφαιρικό του πλαίσιο τη συμφωνία αυτή. Εμείς θέλουμε να ε, βάζουμε όλο και πιο ψηλά τον πύχη προστασίας του περιβάλλοντος, ώστε να ζουν οι πολίτες μας σε ένα ε, περιβάλλον υγιές. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, όχι μόνο δημιουργήθηκε Υπουργείο Περιβάλλοντος εδώ και τρία χρόνια, αλλά και οργανισμός εποπτείας βελτιώθηκαν τα στάνταρ ποιοτικών ελέγχων και γενικότερα πρέπει να πω ότι υπάρχει μια σειρά μέτρων για την βελτίωση των μέτρων που λαμβάνονται για την προσθήκη του περιβάλλοντος. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των διαφόρων διαφωνιών που προκύπτουν. Είναι φυσικό σε κάθε κοινωνία και για μας, για την κυβέρνηση, είναι αυτό ευκαιρία να προχωρήσουμε. Το θέμα του νερού είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Αναγνωρίζουμε ότι είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα η πρόσβαση στο πόσιμο είδος και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε από τα πλαίσια ε, της διακομματικής εθνικής συμφωνίας να υπάρξει συμφωνία μεταξύ όλων όσον αφορά την υδροδότηση και το πόσιμο νερό. Είναι βασικό δικαίωμα και η κυβέρνηση να λάβει δεσμεύσει για να το εξασφαλίσει σε όλου. Ευχαριστώ. Ο πρώτος ομιλητή ξέχασα να πω, ο πρώτος ομιλητή από την αντιπροσωπεία του Περού, ο Χωσέ Λουι Σίλβα, είναι πρόεδρος εμπορίου και τουρισμού. Α περάσουμε τώρα τον Αντιπρόεδρο Γκαρσάν της Κολομβίας. Ε, και πάλι έχετε πέντε λεπτά στη διάθεσή σας. Ε, αν θέλετε μπορείτε βέβαια να τα μοιραστείτε με τα υπόλοιπα μέλη της Αντιπροσωπείας της Κολομβίας. Έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να υποβάλω κάποιες προτάσεις για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την όλη διαδικασία έγκρισης της εμπορικής συμφωνίας, αλλά να προχωρήσουμε σε θέματα προστασίας τροπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, καθώς και σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Πρώτη μου πρόταση είναι η εξή. Μεταξύ της κυβέρνησης της Κολομβίας εκπρόσωποι όλων των ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να συνεργαστούν ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν κάνει επενδύσεις στην Κολομβία να αναλάβουν δεσμεύσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωνόματων για κοινωνική ευθύνη, εταιρική κοινωνική ευθύνη, για βέλτιστες εργασιακές πρακτικές και προστασία του περιβάλλοντος. Ως παράδειγμα θα σας πω ότι με όλες τις ε, ελβετικές επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στην Ελβετία, στην, ε, στο, στην Κολομβία, έχουμε υπογράψει μία συμφωνία για θέματα προστασίας των, ε, των πολιτών. Άλλο παράδειγμα. Η πολυεθνική Καρφούρ ζήτησε από την ε, ε, Εθνική Σχολή ε, που διαθέτουμε να την βοηθήσει για εργασιακή σχολή που διαθέτουμε να τη βοηθήσει για να δημιουργήσουν συνδικαλιστικά όργανα. Αυτά είναι παραδείγματα ώστε να μπορέσουν και άλλες εταιρείες πολυεθνικές που βρίσκονται στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες να κάνει το ίδιο. Δεύτερη πρόταση και επωφελούμε όχι μόνο εκπρόσωποι της κυβέρνησης αλλά και εκπρόσωποι των ε, συνδικάτων της Αμερικής προτείνουμε στον ΔΟΕ να παρασκευάσει ένα πρόγραμμα μόνιμο ώστε να γίνεται παρακολούθηση των εμπορικών συμφωνιών που συνάπτονται όσον αφορά τη συνδικαλιστική ελευθερία, την εργασιακή ελευθερία και τα δικαιώματα των επιχειρηματιών. Τρίτη πρόταση. Η διαδικασία της απόδοσης στους ιδιοκτήτες των ε, γεών είναι μια δύσκολη διαδικασία, διότι δύσκολα μπορείς να, να πάρει τις γεές που έχουν καταπατηθεί από τις ένομλες παράνομες δυνάμεις και να τη δώσει και πάλι στους αγρότες. Προσπαθούμε, αλλά εάν δοθεί ένα εκτάριο ή ένα στρέμμα ή δέκα μέτρα λιγότερο ή περισσότερο, δεν έχει σημασία αυτό. Που έχει σημασία είναι ότι θέλουμε να δώσουν ως κυβέρνηση πίσω τις γέες αυτούς που τη δικαιούνται και από αυτούς που την ε, πήραν παράνομα. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του προγράμματος θα θέλαμε να δημιουργεί μια ομάδα στην οποία η οποία θα ασχοληθεί και με θέματα ε, αποζημιών που θα δοθούν σε θύματα άλλων αδικιών και συνδικαλιστικών αδικιών και βίας. Για να επιτύχουμε, είτε να αποτύχουμε θα είναι μεγάλη αποτυχία. Τώρα, όλα αυτά τα οποία συζητούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να το κάνουμε στα πλαίσια αυτών των δράσεων που αναλαμβάνει στα πλαίσια της πράσινης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο ΙΕ του χρόνου εμείς έχουμε να κάνουμε απόδοση δεινών κατά κάποιο τρόπο και θα περάσουμε δημόσιες εξετάσεις. Όλες οι κυβερνήσεις θα μπορούν να δουν ακριβώς τι έχουμε κάνει σε θέματα προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων από αυτά τα οποία είπαμε εμείς τι έχουμε ολοκληρώσει, τι έχουμε υλοποιήσει και τι όχι. Είναι σαν να δίνουμε εξετάσεις στο δημόσιο. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τι γίνεται και να συμμετάσχετε εσείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε θέματα λοιπόν ευθροπίνων δικαιωμάτων για φέτος το Δεκέμβριο έχουμε συγκαλέσει μία διάσκεψη την οποία συγκάλεσε η κυβέρνησή μας οι, ομοσ... ομοσπονδίες δημάρχων, οι δικαστικές αρχές και άλλες ερετές αρχές, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, ενώσεις ε, επαγγελματιών, ενώσεις ε, εργαζομένων στην Ήπεδρο, γυναικείες οργανώσεις, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ ε, υπό την ε, ε, αιγίδα επίσης ε, ανωτά των οργάνων που εκπροσωπούνται στα Ηνωμένα Έθνη για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με το θέμα της πρόσφασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οτιδήποτε κάνουμε λοιπόν δεν το κάνουμε σε μια χώρα που ζει σε κλίμα ειρήνης. Εμείς πρέπει να πω ότι έχουμε προχωρήσει τον αγώνα μας κατά των ενόπλων παράνομων δυνάμεων, αλλά ακόμη δεν είμαστε μία χώρα σε κλίμα ειρήνης. Κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε προβλήματα βίας. Σήμερα δολοφονήθηκαν περισσότεροι από πέντε στρατιώτες και αστυνόμοι. Και συνελήφθησαν από τις παράνομες δυνάμεις 11 εργαζόμενοι στην ε, πετρελαϊκό τομέα. Ευχαριστώ. Thank you, Chairman. Ε, Ευχαριστώ. Αρχικά για το ερώτημα του κυρίου Ζαντό για τα τοξικά προϊόντα. Νομίζω ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά ζητήματα. Αφενός ε, έχουμε όλα αυτά που συμφωνήθηκαν για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και μετά έχουμε και την ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων ε, στην Ευρώπη ε, που αποτελούν ζητήματα αρμοδιότητας του κυρίου Μπαγνή. Και σύμφωνα με την συμφωνία, της σύμβαση ελεύθερου εμπορίου, τα προϊόντα που φτάνουν σε εμά από την Λατινική Αμερική την χάνουν τις ίδιες μεταχείρισεις με τα ευρωπαϊκά. Ισχύουν δηλαδή οι ίδιοι κανόνες με τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Νομίζω ότι ρυθμίζεται επαρκώς αυτό το θέμα. Αν υπάρχει πρόβλημα, τότε υπάρχει πρόβλημα με την ευρωπαϊκή ρύθμιση. Όχι με τα συγκεκριμένα προϊόντα που προέρχονται από τη Λατινική Αμερική, τα οποία πληρούν τα ευρωπαϊκά κριτήρια και τις ευρωπαϊκές απαιτήσει. Τώρα, για το ερώτημα του κυρίου Σόλτ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι εύκολο αυτό το κεφάλαιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο εμπόριο. Είναι σίγουρο όμως ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, μπορούν να επιβιώσουν μόνο μέσα σε ένα ε, σταθερό νομικό περιβάλλον. Και αυτό ακριβώς παρέχει η εν λόγω συμφωνία. Αν λοιπόν ε, θέλει μια μικρομεσαία επιχειρήση να επιβιώσει μακροπρόθεσμα, τότε θα πρέπει να διαθέτει ένα ε, σταθερό και σίγουρο πλαίσιο. Αυτό θα παράσχει, θα παράσχει και η ε, συμφωνία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις ευρωπαϊκές και της Κολομβίας και του Περού. Ο κύριο Αλάιζα πρότεινε να επαναδιαπραγματευτούμε την ε, συμφωνία. Θα ήθελα να απαντήσω αλληγορικά, λέγοντας ότι εντελώ θεωρητικά, αν υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση τη συμφωνία, όταν ε, καταλήξουμε στη νέα συμφωνία και πάλι θα έχει αλλάξει η οικονομική κατάσταση. Το νόημα μια τέτοια συμφωνία είναι ότι ισχύει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ορισμένε δεκαετίε. Εντάξει, δεν γίνεται κάθε φορά να επαναδιαπραγματευόμαστε τέτοιε συμφωνίε και εξάλλου δεν βλέπω πώ η οικονομική κρίση ε, θα επηρεάσει τη συμφωνία από την πλευρά της Λατινικής Αμερικής. Αν δείτε τις εξαγωγές που θα κάνουν αυτές οι χώρες προς την Ευρώπη δεν επηρεάζονται καθόλου από την οικονομική κρίση η οποία έτσι καλλιώς δεν είναι και τόσο έντονη αυτή τη στιγμή. Κάνουμε λόγο για ήπια ύφεση, αλλά φαγητό έχουμε ακόμα να φάμε, οπότε εντάξει. Κύριε Σαλαφράγκα, γιατί παίρνει δύο χρόνια, ρωτήσατε. Ενδιαφέρον ερώτημα. και δεν αφορά μόνο αυτή τη συμφωνία. Αυτή η περίοδος πράγματι είναι ιδιαίτερα μακρά και υπάρχουν αρκετοί λόγοι γι' αυτό. Ίσως το Κοινοβούλιο να μπορούσε να δει πώς μπορεί να επιλύσει αυτό το πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα, κατά τη σύναυση μιας συμφωνίας, πρέπει να εξεταστεί από νομική πλευρά. Και αυτό είναι δύσκολο, γιατί ε, το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων δεν είναι ένα οριστικό κείμενο. Κάποιες παράγραφοι πρέπει να αναδιατυπωθούν. Υπάρχουν κάποια, ε, κάποιες εργασίες πρέπει να γίνουν ακόμα. Εργασίες όμως απαραίτητες και για την ε, υλοποίηση στη συνέχεια. Κατά δεύτερον όμως πρέπει να μεταφραστεί σε 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια τέτοια συμφωνία πολύ εύκολα περιλαμβάνει από 1.000 έως και 2.000 σελίδες. Φανταστείτε αν αυτό πρέπει να μεταφραστεί σε 23 γλώσσες. Παίρνει μήνες αυτή η διαδικασία. Ίσως και το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να σκεφτεί μήπως κατά τη διαδικασία, να μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία κύρωσης πριν, ε, ε, πριν την ολοκλήρωση της μεταφραστικής διαδικασίας. Ε, εφόσον πρόκειται για ιδιαίτερα τεχνικά ζητήματα που κανένας εδώ πέρα θα τα διαβάσει. Εσείς, ας πούμε, θα τα διαβάσετε. Εγώ δεν γράφω τίποτα, να ξέρετε. Είναι όμως ε, τεχνικά ζητήματα τα οποία ως αποδέκτη έχουν τις ελληνικέ αρχές. Ε, ούτε εσεί το χρειάζεστε ε, για να το κυρώσετε, γιατί δεν αλλάζει κάτι στο πολιτικό πλαίσιο της συμφωνία. Ίσως λοιπόν θα ήταν καλό το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο και την Επιτροπή να σκεφτούν πώς θα μπορούσαν να διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία τη μετάφραση. Γιατί αυτό είναι ο μόνο λόγο που παίρνει τόσο χρόνο. Ξέ, ούτε σε μένα μου φαίνεται λογικό. Και μετά για την κατασκοπία. Πού είναι η κατάσκοπη, για να δω. Το ελέγξαμε και με τις δικές μας μυστικές υπηρεσίες. η συγκεκριμένη υπηρεσία που λέγεται DAS, ένας ένας υπεύθυνος, δύο ε, έχουν εξοριστεί και 40 αποτελούν αντικείμενο έρευνας και μετά ποιο είναι ακριβώς το όνομα της υπηρεσίας. είναι κάποιο είδους μυστική υπηρεσία. Έχει κλείσει από τον κύριο Δοσάντος, τον πρόεδρο. Και το μόνο που λέει το Γραφείο των Εθνών είναι ότι υπάρχουν εκθέσεις για κατασκοπία, αλλά δεν επιβεβαιώνονται. Το σημαντικό είναι ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία όμως έχει κλείσει. Έχει σταματήσει το έργο της ο επικεφαλής της είναι στη φυλακή, άλλοι έχουν εξοριστεί και 40 υπόκεινται σε έρευνα. Αυτό δείχνει ότι έχουν ε, γίνει βήματα για, αυτό, αυτή την υπηρεσία, την DAS. Δεν ξέρω αν ε, απάντησα στο ερώτημά σας. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο εισηγητής, ε, Δαβίδ, από το ΕΛΚ. E Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους συμμετέχοντες για την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και χρήσιμη ε, συζήτηση για να μπορέσουμε και εμείς να αποφασίσουμε. Νομίζω ότι ε, και στα δύο κογκρέσα θα υπάρξει μια ε, παρόμοια συζήτηση στο επόμενο διάστημα και αυτό θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Το ΕΛΚ θα συμμετάσχει εκεί πέρα και δεν θέλει να ε, λαμβάνει από δεύτερο χέρι τις ε, πληροφορίες. Εγώ λοιπόν παρακολουθούσα εκ του ε, τη διαδικασία και ήμουν ενήμερος. Κάποιοι συνάδελφοι ε, λυπούνται που δεν συμμετέχουν και οι τέσσερις χώρες ε, της κοινότητας των Άνδεων σε αυτή την συμφωνία. Το Εκουαδόρ και η Βολιβία εψήφισαν στην Ολομέλεια των Εθνών για τη Συρία 12 κατά και οι δύο ήταν από, τις, από χώρες των Άνδεων. Επομένως, Επίτροπε, σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση του Εκουαδόρ το Δεκέμβριο, παρακαλώ να έχετε κατά νου και αυτή την πολιτική πτυχή που έχει νόημα εδώ. Μπορούμε πολλά να αντλήσουμε από τα όσα είπε ο εκπρόσωπος ε, του ΔΟ εδώ. Ε, τα, τα κύρια στοιχεία των διαπραγματεύσεων είναι τα κοινωνικά, εργασιακά και δημοκρατικά δικαιώματα. Ε, επιτρέψτε μου να στείλω και την ε, τελευταία έκθεση του Human Rights Watch, που είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη οργάνωση. Παρακαλώ, διαβάστε το κεφάλαιο για την βία και τις δολοφονίες συνδικαλιστών στην Κολομβία. Μπορώ να σας τη στείλω, άμα θέλετε η Κολομβία και το Περού έχουν υπογράψει όλε τι συμβάσει ε, του ΔΟΑ και αυτό είναι πολύ θετικό. Τώρα για την ΕΤΟΚ, ε, την TUCA μάλλον, υπάρχει εδώ μια διαφορά. Υπάρχουν δημόσια, ε, υπάρχουν δηλαδή συνδικάτα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Τι γίνεται όμως με τις δεσμεύσεις των δύο αντιπροέδρων. Εκπροσωπούν δύο κυβερνήσεις από δύο διαφορετικούς πολιτικούς πόλους. Και ε, παρόλα αυτά έχουν την ίδια άποψη σε ό,τι αφορά την ε, Συμφωνία Ελεύθερο Εμπορίου, ότι μπορεί να βοηθήσει αυτή η συμφωνία την υλοποίηση όλων των νομικών ε, διατάξεων που υιοθετούνται ε, στι χώρε σα και θα εφαρμοστούν. Ένα άλλο θέμα του εκδημοκρατισμού και όλων των ε, διαδικασιών, όπως προβλέπετε από την ε, κοινωνία των πολίτων και οι δύο εκπρόσωποι μας έδωσαν την δυνατότητα να καταλάβουμε ότι έχουν μάτια και αυτιά ανοιχτά και βλέπουν οποιοδήποτε λάθος. Και τελικά θα ήθελα να κάνω αναφορά στην παρέμβαση του Επιτρόπου Ντεκούχ που μίλησε για την εγγύηση αμοιβαίων ωφελών και για τα δύο μέρη. Όλες οι μελέτες λέγουν ότι τα ΑΕΠ των χωρών αυτών μετά από την σύναψη της εμπορικής συμφωνίας θα αυξηθούν. Ξέρουμε κάθε ε, χρόνο ότι υπάρχουν, ε, ε, υπάρχει βελτίωση του ΑΕΠ. Θα ήθελα λοιπόν να το μελετήσουμε το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε να κάνουμε τώρα με μια πολιτική απόφαση που πρέπει να ληφθεί και κρίνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να επομιστεί την ευθύνη που του αναλογεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φτάνουμε στο τέλος ε, μιας ε, μακροσκελέστατης ανταλλαγής απόψεων. Χαίρομαι που είχαμε μια τόσο ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση με συμμετοχή εκπροσώπων και τρίτων χωρών. Νομίζω ότι ερχόμαστε πρώτοι σε αυτό το τομέα και είμαι περήφανος που είμαι μέλος του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ.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 Θα κάνουμε δύο λεπτά διάλειμμα. Θα κάνουμε διάλειμμα για να προετοιμαστούμε για το επόμενο θέμα.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 less than 2%, crucial and important for GSP. Let's resume our proceeding. Ας προχωρήσουμε. Περνούμε στο σημείο 13 της ημέρας της διάταξης. Έχουμε το πρόσθετο πρωτόκολλο για την Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ. για συμφωνία σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την αποδοχή βιομηχανικών προϊόντων, γνωστή και ως ACA, ACAA. Αυτή η Επιτροπή πέρυσι αποφάσισε να ελέγξει την ε, συμμόρφωση αυτής της οδηγίας με την συνολική εξωτερική δράση της Ένωσης απέναντι ε, στο Ισραήλ. Αποφασίσαμε δύο στοιχεία. Πρώτον, να ζητήσουμε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για μια γνωμοδότηση για αυτό το ζήτημα και να ζητήσουμε από την Επιτροπή να έρθει, την Κομισιόν να έρθει στην Επιτροπή μας και να μας ενημερώσει γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα. Δηλαδή, αυτή η συμφωνία που αποτελεί αναβάθμιση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ, αυτή η συμφωνία λοιπόν συνάδει με την εξωτερική πολιτική της Ένωσης ενώπιον του Ισραήλ. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί πριν ε, ψηφίσουμε ε, για αυτή τη διαδικασία. Η ΑΦΕΤ, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, δεν έχει ακόμα παρουσιάσει τη γνωμοδότησή τη. Ε, κοντεύουν όμω. Και ο Επίτροπος Δε Γιούχτ θα μας ε, μιλήσει εκ μέρους ε, της Κομισιόν για αυτό ακριβώς το ζήτημα. Εφόσον είμαι εξοφίσιο εισηγητής για αυτή τη συμφωνία, θα αναφέρω στα ζητήματα τα οποία θα θέλαμε να απαντηθούν. Αυτό το ζήτημα πολιτικής συνοχής ε, είναι κάτι το οποίο το εξέτασε η Επιτροπή και ποια είναι η αίσθηση της Επιτροπής από αυτού. Πιστεύει λοιπόν η Επιτροπή ότι η αναβάθμιση των εμπορικών σχέσεων με το Ισραήλ δεν αντιβαίνει στις θέσεις της Ένωσης ε, σχετικά με το Ισραήλ. Ιδιαίτερα την ειρηνευτική διαδικασία, την θέση του Ισραήλ απέναντι στην Γάζα, τους επικισμούς και όλα αυτά. Εμπόδια Ε, στην ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ του κράτου Ισραήλ και τη Παλαιστινιακή Αρχή. Όλα αυτά θα θέλαμε να απαντηθούν. Δίνω λοιπόν το λόγο απευθεία στον Επίτροπο του Χιούχτ και στη συνέχεια θα έχουμε σύντομη ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής και τον Επίτροπο. Παρακαλώ. Thank you. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. η σύνδεσή μας, με το Ισραήλ είναι πολύ σημαντική και πολύ τιμή και για τις δύο πλευρές. Και στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής ε, Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ και με την ε, συνέχιση του σχεδίου δράσης ε, για την πολιτική καλής γειτονίας που υιοθετήθηκε το 2005. Αυτό δεν είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε πρόσφατα. Πρέπει να πάμε πίσω 10 χρόνια στην ε, συνεδρίαση Euromed στο Τολέδο. Τότε λοιπόν ένα σχέδιο δράσης για την ε, διευκόλυνση του εμπορίου και των επενδύσεων ενεργοποιήθηκε και μετά είχαμε και την ε, συνεδρίαση στο Παλέρμο το οποίο οδήγησε σε εντατικές εργασίες ε, με τους ε, Ισραηλινούς εταίρους και είχαμε και διαδικασία αξιολόγηση συμμόρφωσης. Το Ισραήλ είναι μία από τις χώρες στην περιφέρεια που, δείχνουν, που δείχνει να ενδιαφέρεται να συμμορφωθεί ε, με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή εξετάζουμε το ενδεχόμενο να επιταχύνουμε την προπαρασκευή για τις διαπραγματεύσεις ΑΚΑ για να ξεκινήσουν στο άμεσο μέλλον. Υπό αυτή την πολιτική λοιπόν και το σχέδιο δράση που υιοθετήθηκε το 2005 δεσμεύτηκαν και οι δύο εταίροι ε, να επιταχύνουν τη δικασία για την ε, μελλοντική ε, συμμόρφωση και αποδοχή των βιομηχανικών προϊόντων, τη λεγόμενη ΆΚΑ. Πέντε χρόνια μετά, το Μάιο του 2010, το Συμβούλιο υπέγραψε την Συμφωνία ΆΚΑ και πάλι θα ήθελα να ξαναπώ ότι είχαμε τη φιλοδοξία να επεκταθεί η ΆΚΑ ε, σε πάνω από μία χώρες. Πράγματι στο σχέδιο δράσης 2004-2005 είχαμε και με το Μαρόκο και την Τινησία με παρόμοιες διατάξεις και έτσι άκαμε με το Ισραήλ δεν αποτελεί ιδιαίτερο προνόμιο, εντάσσεται στο πλαίσιο των, των υφιστάμενων εμπορικών μας ε, σχέσεων ε, με χώρες όχι μόνο αυτής της περιοχής αλλά και με τις Ασίας και αλλού. Οι διαδικασίες, οι ξεκίνησαν μόλις το 2008 όταν το σχέδιο δράσης του 2005 σχεδόν είχε ε, εκπνεύσει. Όλα αυτά βέβαια είναι ανεξάρτητη συζήτηση από την αναβάθμιση. Δηλαδή η δέσμευση ε, για την ε, συμφωνία ΑΚΑ προηγείται ημερολιακή χρονικά και δεν συνδέεται με την δέσμευση αναβάθμισης. Το σχέδιο δράσης παρέμεινε το έγγραφο αναφοράς για την διαδικασία αυτή και η προσέγγιση υλοποιήθηκε αυστηρά και συνεχίσαμε ε, στο ίδιο πλαίσιο, δηλαδή με το σχέδιο δράση 2005. Τώρα δεν θέλω να εξηγήσω τι είναι μια τέτοια συμφωνία. Άκα. Βεβαίως και το γνωρίζετε, αλλά θέλω να το επαναλάβω είναι μια ε, εμπορική συμφωνία που θέλει να άρει εμπόδια στο εμπόριο και στα βιομηχανικά προϊόντα. Αποτελεί συμφωνία αμοιβαία αναγνώριση και έτσι ε, συμφωνούμε ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση τα Ισραηλινά φαρμακευτικά προϊόντα ε, παρασκευάζονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στην πράξη, όλα τα, τα προϊόντα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς ε, άλλη διαδικασία. Τα ωφέλη είναι ότι οι οικονομικοί φορεί και στι δύο πλευρές ε, εξοικονομούν χρόνο και χρήμα. Και οι Ευρωπαίοι και οι Ισραηλινοί καταναλωτές ε, έχουν ωφέλη σε, σε επίπεδο κόστους. Έτσι έρουμε τα, τα εμπορικά εμπόδια. Προς το παρόν έχουμε έναν τομέα που ε, εμπλέκεται, το, το τομέα της φαρμακοβιομηχανίας. Το Ισραήλ λοιπόν ε, έχει συμμορφωθεί με την νομοθεσία και βεβαίω όλε αυτέ τι πληροφορίε πρέπει να τι βρείτε στο παράρτημα του, του κειμένου ε, που έχει, δοθεί στο Κοινοβούλιο. Λοιπόν, σύμφωνα με την ΆΚΑ υπαγόμαστε στο άρθρο 83 της Συμφωνίας Σύνδεσης ε, ε, και σε επίπεδο επικράτειας δεν ε, δεν περιλαμβάνονται τα εδάφη που περιήλθαν στην επικράτεια του Ισραήλ μετά το 1967. Θα ήθελα να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να τονίσω το πλαίσιο ενός δομημένου διαλόγου αρκετά ζητήματα τα οποία θα μα απασχολήσουν στη συνέχεια. Η συνεργασία και ο συντονισμό ε, σε ορισμένου τομεί. Νομίζω ότι η Επιτροπή θα είναι σε θέση να παρουσιάσει σε εσά και στο Συμβούλιο μια πρόταση για το σχέδιο πρόσβαση στην αγορά μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Ελπίζω επίσης να υποβάλω την πρόταση μόλις έχουμε ε, το, ε, το, κείμενο για τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ Όλα αυτά για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τους εταίρους μας και, την, ε, το σεβασμό των ε, δικαιωμάτων. Ε, βεβαίως και θα υποβληθεί σε εσά και στο Συμβούλιο για την χρηματοπιστωτική ευθύνη του πιστωτή. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξυγχρονίσουμε τα εμπορικά μέσα με την διεύρυνση και ενίσχυση των διαβουλεύσεων. Ε, οποιαδήποτε ε, πρόταση θα γίνει ε, το 2013. Προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Έχουν ζητήσει πάρα πολύ το λόγο και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βάλω το ρολόι για να αρχίσει να μετράει και θα δώσω στον κάθε ένα ομιλητή δύο λεπτά. Ας ξεκινήσουμε με την Λουσία Αντρίκινεν που είναι ε, σκιώδηση από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ε, θα ήθελα να καλωσορίσω την ε, πρόοδο που έχει επιτευχθεί και επιτρέψτε μου για άλλη μια φορά να υπογραμμίσω ότι αυτή είναι μια συμφωνία ε, που αφορά αμοιβαίως αποδεκτά ε, αμοιβαίες αποδεκτές προδιαγραφές στα φαρμακευτικά προϊόντα. Όμως, ε, εάν δεν προχωράμε στο θέμα αυτό, κρατάμε όμοιρο τη δική μας την φαρμακευτική βιομηχανία. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί στη τελική ανάλυση πρόκειται για φάρμακα και δεν πρόκειται για όπλα. Από την ε, Βερονίκ Ντεκάιζερ, η οποία είναι η εισηγήτρια στο θέμα αυτό, προτάθηκε να συσταθεί μια ενδιάμεση έκθεση και θα ήθελα να ζητήσω από τον Επίτροπο κ. Ντεπούχτ το εξή ε, κατά πόσον μπορεί να υπάρξει μια νέα συζήτηση διαπραγματεύσεων Αλλιώς ε, θα υπάρξουν νέες καθυστερήσεις σε αυτή τη συμφωνία ΆΚΑ. Και τέλος ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά την ε, διαφωνία που υπάρχει της λόγω νομοθεσίας με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ανταλλαγή φαρμάκων. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα ήθελα να ενθαρρύνω τους συναδέλφους να σκεφτούν πάνω στο θέμα αυτό. Υπό την προπόθεση βέβαια θα υπάρχει το στομό των δυνατών η συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, ε, να ακούσουμε καταρχήν ε, το θέμα της ε, συνέπειας της συμφωνίας σχετικά με την συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ισραήλ. Εμείς καλύτερα να μην εμπλακούμε στις δικές τους τις συζητήσεις. Μαρίτια Σάκε από την Ομάδα των Φιλελευθέρων. Επόμενο μιλήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε πίτροπε. Θα είμαι πάρα πολύ ε, σύντομη, δεν θα χρειαστώ ούτε καν δύο λεπτά. Η δική μας η πολιτική ομάδα θα ήθελε να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για αυτό το πρωτόκολλο SDSA. Και για μας ε, να σας πω ότι ε, αυτό δεν εμπίπτει στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για εμά τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά δεν εμπίπτει εδώ το θέμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ε, θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε ξεχωριστά από τα ανθρώπινα δικαιώματα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ε, πρόεδρος, υπάρχει ήδη ένα χρονοδιάγραμμα από το κ. Βαϊβέρε, από η κυρία Βαϊβέρε, από το ΕΛΚ. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι προφανές ε, ότι οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παραγωγή θα ωφεληθούν από αυτή τη συμφωνία. Ε, και θα συμβεί αυτό διότι το Ισραήλ έχει μονόπλευρα εφαρμόσει την ε, συμφωνία αυτή ε, στο πλαίσιο των διμερών υποχρεώσεων. Να πω τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση το εξή. Οι Ευρωπαίοι ασθενεί θα επωφεληθούν από ένα ευρύτερο φάσμα ιατρικών προϊόντων γιατί δεν θα υπάρχουν οι προϋποθέσεις συμβατότητας. Δεύτερον, οι ε, εξαγωγείς φαρμακευτικών προϊόντων θα ε, επωφεληθούν και αυτοί από τότε δεν θα υπάρχει τόσο προσεκτισμό, θα περιστούν τα χρονικά περιθώρια και τρίτον, οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτές θα επωφεληθούν εξοικονομώντας χρόνο και σεβόμενες τις εισαγωγές του Ισραήλ. Ε, δυστυχώς έχει γίνει λανθασμένα μια συμφωνία για αναβάθμιση των σχέσεων Ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ κατ' ουσίαν η συμφωνία αυτή μπαίνει ε, στη συμφωνία που ήδη υπάρχει στο πλαίσιο της διαδικασίας της Βαρκελόνης. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν υπάρχει λόγος να πολιτικοποιούμε αυτή τη συμφωνία ή να τη συνδέουμε με άλλα θέματα. Ανταυτού θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις ε, θετικές ε, επιπτώσεις και για τις δύο πλευρές και θα έλεγα ότι δεν πρέπει να καθυστερούμε πλέον όσον αφορά τη συμφωνία αυτή, να της δώσουμε πράσινο φως. Πολύ ωραία, λέει ο Η κυρία Λατφόρτ, ε, που δεν είναι μέλος αυτής της Επιτροπής, αλλά σας καλωσορίζουμε παρόλα αυτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω για το θέμα αυτό. Και εγώ χαίρομαι που ε, σημειώνουμε πρόοδο, διότι νομίζω ότι έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από τότε που ορίστηκε ο πρώτος εισηγητής. Και Αυτό μάλλον είναι και ρεκόρ βραδύτητας. Το πρώτο που θέλω να πω είναι το εξής. Πρέπει να προχωρήσουμε το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να προβεί σε δημοκρατική επιλογή όσον αφορά στην έγκριση ή απόρριψη αυτής της ε, συμφωνίας. Η δική μου θέση είναι ότι πρέπει να εγκριθεί η συμφωνία. Αλλά Νομίζω ότι είναι αντιδημοκρατικό να μην πάει το θέμα στην Ολομέλεια μετά από δύο ολόκληρα χρόνια. Ε, πρέπει λοιπόν ε, πάση θυσία να ληφθεί πλέον μία απόφαση. Και όπως είπαν και άλλοι, ε, εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξουν πρακτικά πλεονεκτήματα, όχι μόνο για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, αλλά και για τους Ευρωπαίους εξαγωγής προς το Ισραήλ. Ε, μια συμφωνία η οποία θα περιορίζει τη γραφειοκρατία στις ε, εισαγωγές, εξαγωγές ε, φαρμακευτικών προϊόντων. Σε περίοδο λιτότητας νομίζω ότι είναι ευπρόσδεκτη η πιθανή μείωση των δαπανών για την υγεία. Και τρίτον, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίσως αυτό μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες παρεμφερείς συμφωνίες. Την Ισία, ίσως η Ορδανία, Μαρόκο να ακολουθήσουν και αυτές. Εάν λοιπόν καθυστερήσουμε κι άλλο, τότε τι μήνυμα θα περάσουμε σε αυτές τις χώρες για, για ίδια μέτρα και ίδια σταθμά. Ε, δεν με πέρυσι την συμφωνία με την Παλαιστίνη για γεωργικά και αλληλευτικά προϊόντα. Κατόπιν τούτου όπως ε, ε, μόλις τώρα είπε και η συνάδελφός μου, προφανώς και μας ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά όταν μιλάμε για εμπόριο, μιλάμε για τεχνικά θέματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούμε να τα εξετάσουμε σε πολιτικό πλαίσιο, ακόμα και σε στενότερο διάλογο με τους ε, συνομιλητές μας, προσπαθώντας να τους προσετεριστούμε. Εδώ είμαστε για να συζητάμε για την πολιτική συνέπεια και όχι για τα οικονομικά ωφέλη μιας συμφωνίας. Δηλαδή, εδώ βρισκόμαστε να μιλάμε για πολιτικά θέματα και όχι εμπορικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, αν αυτό, αυτή είναι η ουσία του θέματος, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ε, μια ψηφορία για την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας δεν θα έχει πολιτικές ε, προεκτάσεις. Προφανώς θα υπάρξει προστιθέμενη αξία εμπορικά αλλά και πολιτικά θα υπάρξουν προεκτάσεις. Θα εκπέμψουμε σαφέστατο μήνυμα πολιτικό μήνυμα προς αυτή την περιοχή, όχι μόνο στο Ισραήλ, αλλά και στις όμορες χώρες. Ε, και αυτές ε, πρέπει να δουν ότι είμαστε συνεπείς ε, όσον αφορά την εμπορική πολιτική που ακολουθούμε και την εξωτερική. Γι' αυτό λοιπόν κάνω την εξή ερώτηση προς την Κομισιόν και προς όλους μας. Σε σχέση με ένα ή μάλλον δύο χρόνια παλαιότερα, η κατάσταση επιτόπου άλλαξε προς το καλύτερο. Δηλαδή, σημειώθηκε πρόοδος σε, σε επίπεδο ειρηνευτικής διαδικασίας ή όσον αφορά τον πλήρη κατάλογο. Δεν έχει τώρα νόημα να επαναλαμβάνουμε τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Ισραήλ, αλλά και προς, ούς, προς πολλούς άλλους ε, παίκτες της περιοχής. Αν αυτό είναι το θέμα που συζητάμε, νομίζω πρώτα απ' όλα πρέπει να περιμένουμε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων που ε, την επεξεργάζονται. Δεν ξέρω αν έχουν ψηφίσει ήδη επ' αυτής. Νομίζω πως όχι. Ε, πρέπει να είμαστε συνεπείς ε, και με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων όσον αφορά το θέμα αυτό. Η δική μου η άποψη είναι ότι θα ήταν αφελές να λέμε ότι πρόκειται εδώ απλά και μόνο για ένα εμπορική φύσεως θέμα χωρίς ε, πολιτικές ε, προεκτάσεις. Η κυρία Βερονίκ Ντεκάιζερ δεν είναι μέλος αυτής της Επιτροπής, είναι όμως των εξωτερικών υποθέσεων. Ίσως λοιπόν μπορεί να μας ενημερώσει για τις ε, διαδικασίες που ακολουθούνται στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Ε, είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Και υπάρχει έγγραφο και αίτηση νομικής ε, γνωμοδότησης. Όλα αυτά είναι εν εξελίξη. Τώρα, θα ήθελα να σας πω ότι εμένα όλα αυτά τα οποία ακούμε εκπλήσουν κάπως, διότι βλέπω ότι στην Επιτροπή σας λέτε ότι πρόκειται για τεχνικό φάκελο, για τεχνική συμφωνία. Εάν ε, κάποιος χαιρετίζει την όλη διαδικασία ΆΚΑ γενικά και για το κοινοτικό κεκτημένο, το οποίο θα επιτρέψει αργότερα σε κάποιες άλλες χώρες να απλοποιήσουν διαδικασίες, είμαι εγώ, εάν κάποιος χαίρεται για αυτού του είδους την ε, διαδικασία. Τώρα, ούτε η συνθήκη της Λισαβόνας, ούτε τα κείμενα τα οποία ψηφίσαμε εμείς οι ίδιοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν μπορούν να μας επιτρέψουν να εξετάσουμε χωριστά την πολιτική από την εμπορική διάσταση. Μας λένε πολιτική γυτνίασης. Συν, συ, συν. Δεν θα κάνουμε τίποτε το αρνητικό, αλλά όσοι θέλουν κάτι περισσότερο θα πρέπει επίσης να δώσουν κάτι περισσότερο, ακόμη και σε θέματα πρόσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό υπάρχει με απόλυτη σαφήνεια, έχει λεχθεί ρητό, υπάρχει η συνθήκη τη Λισαβόνα και μου λένε «Μα ονειρεύεστε κυρία Κάιζερ». Δεν ονειρεύομαι, δεν θα έπρεπε να ψηφίσετε. Κύριε Επίτροπε, εδώ τίθεται το θέμα της συνεκτικότητας και της συνέπειας. Μπορούμε να λέμε από τη μια ότι πρόκειται για εμπορικό θέμα και από την άλλη, ναι, ακούστε, ε, τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, είναι πολιτικό θέμα. Θα συζητήσουμε χωριστά στο Συμβούλιο Σύνδεση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ και στην συνάντηση του Φεβρουαρίου πέρσι, το 2011, έθεσε ερωτήματα και έκανε σχόλια πολύ σοβαρά στο Ισραήλ η Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα της Γάζας, τα ανθρώπινα δικαιώματα η κατάσταση όμω για όλα αυτά τα θέματα που θέσαμε τότε επιδεινώθηκε. Αν στα πλαίσια αυτού του διαλόγου δεν επιτυχάνει τίποτα, αλλά όλα είναι πιο αρνητικά, μέσω οποίου μέσου μπορούμε να περιμένουμε μία βελτίωση. Γι' αυτό με εκπλήσει αυτού του είδου η ε, διαδικασία που ακολουθείτε από εσάς. Σκιώδης ηγετής, ο κύριο Σαντό. Χαίρομαι που λέγουν οι συνάδελφοι από το ΕΛΚ που επιτίθενται στις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. Θυμάμαι ε, κάτι το οποίο έχει λεχθεί και θα ήθελα όλοι μαζί να κάνουμε κοινό αγώνα για να μειωθούν οι τιμές των φαρμάκων στην Ευρώπη. Είμαι μαζί τους. Ακούστε, αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε όντως ε, σε βελτίωση της ε, σχέσης από τεχνικής πλευράς, αλλά από πολιτικής πλευράς αυτό είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται. Βλέπουμε τις πολιτικές αποχρώσεις διαφορές. Άκουσα την κυρία Στόνα να λέει συγκεκριμένα πράγματα για την πολιτική και την στρατηγική επικισμού που ακολουθεί το Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες. Λέει, είπε ότι πρόκειται κατά στρατήγηση του διεθνούς δικαίου, είπε ότι τίθεται πρόβλημα και από τη στιγμή κατά την οποία κάνουμε με αυτό το πνεύμα την πολιτική ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η έγκριση ή το ξεπάγωμα του ΆΚΑ αν θέλετε είναι κάτι το οποίο είναι αντιφωσικό σε σχέση με αυτό το οποίο είπε πρόσφατα η Λέιδη Άστον εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. David Martin. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το έργο μου είναι πλέον πιο εύκολο μετά τους τρεις τελευταίους ομιλητές, αλλά με προβλημάτισε αρκετά η αρχή της συζήτησης. Ε, δεν θεωρώ αυτή τη συμφωνία ως αναβάθμιση ε, σε τεχνικό επίπεδο των συμφωνιών ε, με την Ευρώπη, των σχέσεων με την Ευρώπη. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ οικονομικά το Ισραήλ και εφόσον το Ισραήλ συνεχίζει την ε, να τιμωρεί ε, την ε, Γάζα και καταστρατηγεί τα δικαιώματα των πολιτών και των παιδιών στη Γάζα και κλέβει την γη των Παλαιστινίων αγροτών. Πώς γίνεται εμείς να ε, κοινότητα αξιών και από την άλλη να υπογράφουμε την ΆΚΑ. Δεν βγάζει νόημα. Αυτό κάνει το Ισραήλ. Ε, βάζει στην άκρη ε, τη λογική, αλλά εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο. Αυτή η συμφωνία είναι απαράδεκτη στην τρέχουσα κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Μιλάμε για πολιτική συνοχή εδώ πέρα και δεν, μπορούσα να, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τα όσα είπε ο Μάρτιν. Εμείς και με τον Ντέιβιντ ήμασταν στη Γάζα τον Ιούλιο και συνομιλούσαμε με πρόσφυγα με την, ε, με την ε, υπηρεσία προσφύγων ε, των Εθνών είναι μια ε, περιοχή αποκατοχή 49% ανεργία, 39% γεωργικών εκτάσεων υπό απαγόρευση κυκλοφορίας. επισκεφθήκαμε τον Υπουργό Υγείας Πασαμνή, μας είπαν ότι 500 ασθενείς πέθαναν, έχασαν τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια λόγω απώλειας φαρμακευτικών σκευασμάτων. Ε, και είχαν τεράστια έλλειψη ιατρικών σκευασμάτων όπως ε, γάντια για παράδειγμα, ιατρικά γάντια λόγω ε, μόνο του εμπάργου από το Ισραήλ. Και από την άλλη είχαμε τόσα ε, τόσα μηχανήματα τα οποία δεν μπορούσαν να εγκατασταθούν επειδή το Ισραήλ δεν, άφηνε να, να, δεν έδινε πρόσβαση σε τεχνικούς. Είδαμε κτίρια χωρίς ε, ε, να έχουν ολοκληρωθεί. Ο πόλεμος στους Παλαιστινίους συνεχίζεται κάθε μέρα και δεν είναι δυνατόν εμείς ενώπιον όλου του κόσμου όλη τη φιλίου ε, που ζητούν από εμά να ε, βρούμε μια λογική εμπορική ε, πολιτική, ξαφνικά να το ρίξουμε κάτω από το χαλί και να πούμε εντάξει δεν πειράζει, είναι καλό για το εμπόριο, θα φτηνίνουν τα φάρμακα, ενώ στην πράξη καταπιέζονται οι Παλαιστίνοι. Εδώ την προηγούμενη εβδομάδα ε, είπαμε εδώ μάλιστα στο Κοινοβούλιο ότι είναι, παράνομη η έπικοι. Γι' αυτό λοιπόν ε, ζητώ να μην ψηφιστεί τίποτα έω ότου το Ισραήλ καταφέρει να βρει ένα ε, ε φιλήσυχο και ειρηνικό ε, μέλλον για το μέλλον. Κύριε Κασουλίδη, ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Κατά τη γνώμη μου, η συμφωνία ΑΚΑ που εξετάζουμε σήμερα δεν είναι ούτε πολιτική ούτε τεχνική αναβάθμιση των σχέσεών μας με το Ισραήλ. Ο Επίτροπος Δεγκούχτ ήταν ξεκάθαρος, είπε ότι αναβαθμίζει και επικαιροποιεί μάλλον, επικαιροποιεί και δεν αναβαθμίζει βρίσκεται στο πλαίσιο τη ευρωμεσογειακή ε, ε, εταιρική σχέση όπου συνάπτονται ε, εταιρείε σύνδεση, συμφωνίες σύνδεση και όπου όλοι συμμετέχονται ανεξαρτήτω πολιτικών κριτηρίων κλήθηκαν να βελτιώσουν ε, τις ε, συμφωνίες σύνδεσης με πρωτόκολλα σαν αυτό. Ναι, πράγματι θέλουμε more for more, περισσότερα για περισσότερα, όχι more for less, περισσότερα για λιγότερα. Και σίγουρα, εάν θα θα απαρνηθούμε την επιρροή που έχουμε στην Μέση Ανατολή για να ε, επηρεάσουμε την καταστάση στην Μέση Ανατολή. Αν είναι έτσι, δεν συμφωνούμε με την ΆΚΑ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι έχω εκφράσει τις ανησυχίες μου. Ε, φοβάμαι ότι πολλές φορές ε, ε, υφαρπάζουν την άποψή μας ε, για πολιτικής φύσεως θέματα. Διερωτώμε κατά πόσον πράγματι είναι εδώ ο σωστός χώρος για να τεθεί το θέμα αυτό. Έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά για να προωθηθεί το εμπόριο. Το θέμα είναι ότι πράγματι ε, υπάρχουν όλο και περισσότερα προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με διακριτική μεταχείριση. Εγώ είμαι φίλος του Ισραήλ, με κριτικό βέβαια πνεύμα και καταλαβαίνω θέματα όπως είναι επικισμός, ε, οι αποκλεισμοί, αλλά δεν νομίζω ότι εδώ σε αυτήν την Επιτροπή, στην Επιτροπή Διεθνούς Συμπορίου είναι ο κατάλληλος ε, χώρος για να προβληθούν τέτοιου θέματα. Αυτή η συμφωνία είναι σημαντική. Θα φέρει φτηνότερα φάρμακα. Το Ισραήλ είναι μεγάλη φαρμακοπαραγωγός ε, χώρα και θα φέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτηνότερα φάρμακα. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Επίσης, η Κνεσέτ έχει ήδη θεσπίσει νομοθεσία θα ήταν λοιπόν ε, κακό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, θα έβλαπτε την αξιοπιστία της αν δεν ανταποκρινόταν. Όπως και τον Ιανουάριο σας είπα ανησυχώ γιατί κατά κάποιον τρόπο υφαρπάσουν την άποψή μας και από τα πολιτικής φύσεως θέματα μας επιβάλλουν απόψεις σε θέματα που έχουν σχέση με το εμπόριο. Η συμφωνία ΆΚΑ είναι μια τεχνικής φύσεως ε, συμφωνία και ως έχει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ, ε, στις, ε, στα κατεχόμενα, στις υποκατοχήν περιοχές, προφανώς υπάρχουν πολιτικές προεκτάσεις. Αυτό νομίζω είναι απόλυτα σαφές για όλους. Όμως, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η ιδέα ότι η συμφωνία ΆΚΑ πρέπει να αντιμετωπίσετε ως ένα εργαλείο για να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση του Ισραήλ έτσι ώστε να αλλάξει την ε, πολιτική της, αυτό ε, δεν είναι ρεαλιστικό. Αν θέλουμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, οφείλουμε να προτείνουμε ένα σημαντικό, ένα ευρύ πρόγραμμα. Δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να κάνουμε κάτι τέτοιο. Υπάρχει βέβαια πολιτική βούληση για μια τέτοια πρόταση. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε επανέλθει σε αυτό το θέμα. Η συμφωνία αυτή θα πρέπει να στηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. που σημαίνει ότι θα πρέπει να ασκήσουμε θετική πίεση προς την κυβέρνηση του Ισραήλ. Θα πρέπει όμως να χρησιμοποιήσουμε άλλα εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν μπλοκάρουμε αυτή τη συμφωνία, τη συμφωνία ΆΚΑ, νομίζω θα ε, κάνουμε τους εχθρούς του Ισραήλ να αισθάνονται ευχαριστημένοι, αλλά δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα υφίσταται, δεν είναι όμως εδώ ο σωστός χώρος για να λυθεί ε, το πρόβλημα αυτό. Ε, και τελευταίος ο από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα είμαι σύντομος. Κοιτάξτε, εδώ τίθεται θέμα αρχής. Ακολουθούμε πολιτική προσέγγιση. Και βεβαίως και περιμένουμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Συμφωνώ με όλα αυτά που είπαν οι υπόλοιποι προαλήσαντες για το θέμα αυτό. Θέλω όμως να προσθέσω κάτι. Όχι στη Γάζα, αλλά στην ε, Δυτική Όχθη, Όπως έχει πάει στη Δυτική Όχθη και έχει δει το πρόβλημα νερού που υπάρχει, το να μιλάμε εδώ για τεχνικής φύσεως θέματα που έχουν σχέση με τα φάρμακα, Δυστυχώ οδηγεί στο να αγνοούμε τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν άνθρωποι και στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά εδάφη. Γι' αυτό λοιπόν και ω Επιτροπή διεθνού Εμπορίου οφείλουμε το θέμα αυτό να το εντάξουμε μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και να μην τον υποβαθμίζουμε σε τεχνικής φύσεως ε, θέμα. Γιατί ακόμα και τεχνική φύσεως θέματα σε τόσο δύσκολες ε, και αντίξωες συνθήκες που υπάρχουν στη διένεξη Ισραήλ-Παλαιστίνης, ακόμα και αυτά τα τεχνικής φύσης θέματα παίζουν σημαντικό ρόλο. Κύριε Επίτροπε, ε, θέλετε να απαντήσετε στα σχόλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η απάντηση που έδωσα από τεχνική σκοπιά είναι σαφέστατη διότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2009 πρότειναν ε, και παραθέτω ε, το κείμενο που υπάρχει ε, αποτελεί τη νομική βάση χωρίς να υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αναβάθμιση των σχέσεων με το Ισραήλ. Τέλος της παράθεσης. Αυτή την θέση έχουμε ακολουθήσει στο πρόγραμμα δράσης του 2005 συμπεριλαμβανομένη συμπεριλαμβανομένου και του πρωτοκόλου της Συμφωνίας ΑΚΑ. Αυτά είναι τα γεγονότα. Όμως αυτό το θέμα δεν είναι μόνο τεχνικής φύσεως, είναι και θέμα ε, πολιτικής αξιολόγησης. Αυτή λοιπόν την πολιτική αξιολόγηση την αφήνω στη σοφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόεδρος, κατόπιν τούτου εγώ που είμαι συγητής ε, οφείλω να ολοκληρώσω τη συζήτηση. Και πρέπει να σας πω, εγώ δεν πίστηκα. Δεν πίστηκα για το ότι υπάρχει κάποια συνέπεια ανάμεσα στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Ισραήλ και αυτή την εμπορική συμφωνία. Εδώ μιλάμε για μια συμφωνία που θα δώσει τη δυνατότητα σε 100 εκατομμύρια καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική φαρμακευτική βιομηχανία του Ισραήλ. Περί αυτού πρόκειται. Ε, μιλάμε εδώ για μια σημαντική οικονομικά συμφωνία Βεβαίως και θα ωφελήσει το Ισραήλ. Αυτό είναι απόλυτα σαφές για μένα. Και παράλληλα εκπέμπουμε και ένα μήνυμα προς το Ισραήλ και προς τους Παλαιστίνιους ότι δηλαδή καταδικάζουμε καταδικάζουμε την κατάσταση του Ισραήλ Κοιτάξτε, δεν καταδικάζουμε τον αποκλεισμό της Γάζας, ούτε τους επικισμούς, ούτε και την κατοχή και την προσάρτηση της Δυτικής Ιερουσαλήμ ούτε καταδικάζουμε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων που βρίσκονται στο Ισραήλ, που είναι το δικαίωμα ελεύθερη μετακίνηση, ελευθερία απόκτηση γης, ελευθερία απόκτηση πατρίδας. Το δικό μου το πρόβλημα είναι κατά πόσον ε, θα είμαστε συνεπείς ή όχι σε αυτή την πολιτική ή στις πολιτικές την εμπορική και την εξωτερική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν ε, Ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τη γνώμη της. Θα περιμένουμε και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Και τέλος βέβαια <clears throat> θα αποφασίσουμε εμείς. Επειδή ε, εξοφίσιο είμαι εισηγητής, θα κάνω ό,τι αποφασίσει η Επιτροπή μας. Αλλά προφανώς έχω και εγώ δικαίωμα να έχω τη δική μου άποψη. Και νομίζω ότι έτσι μπορούμε και να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Μήπως ε, μπορείτε να μου πείτε διαδικαστικό, διαδικαστικό. Ε, μπορείτε να μου πείτε πότε το θέμα θα πάει στην Ολομέλεια. Το Κοινοβούλιο να μπορεί να αποφασίσει. Ε, συγγνώμη, δεν ξέρω. Μπορείτε να μου πείτε πότε προβλέπετε την ψηφορία στην Ολομέλεια. Ο πρόεδρος δυστυχώς ομιλεί εκτός μικροφώνου. Κοιτάξτε, για τον Ιούνιο προβλέπεται η ψηφορία στην Ολομέλη. Πάμε στο επόμενο θέμα, το 14. Ε, πρόκειται για την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης μίμηση μεταξύ αφενός Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών και αφετέρου άλλων χωρών. Εδώ πρόκειται για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο και ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Ντέβιτ Μάρτιν. Όπως ξέρετε πολύ καλά, αύριο ε, θα έχουμε ένα εργαστήριο που θα ασχοληθεί με ακριβώς αυτό το θέμα. Εγώ λοιπόν προτείνω τα επίμαχα θέματα αυτής της συμφωνίας να τα αφήσουμε για αύριο. Και σήμερα να ασχοληθούμε με τα διαδικαστικά. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι υποχρεούστε να κάνετε αυτά που λέω, μπορείτε να κάνετε και κάτι άλλο. Πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά δέκα λεπτά έχουμε από ό,τι βλέπω για τη συζήτηση. Οι διερμηνείς μου είπαν θα μείνουν άλλα 10 λεπτά. Έχουμε 20-25 λεπτά. Αν έχουμε 20 λεπτά, εγώ πιστεύω ότι το θέμα είναι τόσο περίπλοκο και δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλοι μας μπορούμε να εκφραστούμε μέσα σε 20 λεπτά και να πάρουμε υπεύθυνε απαντήσεις από τον Επίτροπο. Γι' αυτό προτείνω είτε να καθυστερήσουμε σήμερα, όχι για 20, αλλά για πολλή ώρα παραπάνω. Ή να το ε, μεταθέσουμε ε, το θέμα, να το αναβάλουμε για αύριο. Γιατί, κοιτάξτε, 20 λεπτά δεν φτάνουν για αυτό το τόσο ε, περίπλοκο θέμα. Να μας πούν οι συντονιστές ε, την άποψή τους. Πρόεδρε, με συγχωρείτε, έχουμε καθυστερήσει, αλλά να εκμεταλλευτούμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας ε, και αν δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, να διακόψουμε. Αλλά να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί είναι παρόντες. Να δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο του Γιούχ για να κάνει την παρουσίασή του σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα κάνω τώρα την ανακοίνωσή μου, αλλά δεσμεύομαι να είμαι εδώ αύριο και στη συζήτηση. Όποτε και αν συναντηθείτε, εγώ θα, θα τα καταφέρω να έρθω. Εάν διαβάζετε τις, ε, διαβάζετε τις εφημερίδες και βλέπετε τη συζήτηση στο διαδίκτυο, ενδεχομένως να πιστεύετε ότι το, αυτή η συμφωνία σημαίνει το τέλος της δημοκρατίας ε, και τον περιορισμό ε, της πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτικά σκευάσματα σε αναπτυσσόμενες χώρες. Για παράδειγμα, χθε το βράδυ έλαβα 179 email από αυτού. Παρακολουθώ και εγώ αυτό το διάλογο, ακούω προσεκτικά τους ε, πολίτε ε, που βγήκαν στου δρόμου για να εκφράσουν την ανησυχία του για την άκτα. Ε, πολλοί πολίτε σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Κάποιοι από εσά σα πούνε ότι ένα εκατομμύριο μπορεί να κάνουν και λάθο. Αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα νομίζω ότι είναι ευθύνη μα ω πολιτικών να διευκρινίσουμε, ξεκαθαρίσουμε τις παρανοήσεις και να επιλύουμε τέτοια προβλήματα. Πρέπει να ε, εξηγούμε τα, τα στοιχεία, τα δεδομένα, την κατάσταση για να διασκεδάζουμε οποιουσδήποτε φόβους. Νομίζω ότι αυτοί οι φόβοι δεν βασίζονται στην πραγματικότητα. Γι' αυτό το μήνυμά μου προ ε, του Ευρωπαίου πολίτε είναι απλό. Η άκτα δεν ε, αποτελεί επίθεση και απειλή απέναντι στι ελευθερίε σα. Δεν είμαστε στο 1984, είμαστε το 2012, η Άκτα δεν είναι ο μεγάλος αδερφός, ε, είναι μέσω επίλυσης των οικονομικών μας προβλημάτων και το 2012 και μετά. Και το 2012 έχουμε πραγματικά οικονομικά προβλήματα που πρέπει να επιλύσουμε με πρακτικά βήματα και η Άκτα είναι μέρος της λύσης γιατί ε, το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από το κατά πόσο εμείς θα μπορέσουμε να επαναπροσδιορίσουμε τον ε, ρόλο μας σε μια νέα οικονομία. Η δημιουργικότητα και η καινοτομία είναι από τα πιο σημαντικά μας ε, προσόντα και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να σεβόμαστε βεβαίω τα δικαιώματα που υπάρχουν, αλλά πρέπει να δημιουργούμε και νέε θέσει εργασία και οικονομική ανάπτυξη. Αλλιώ δεν έχει νόημα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσά, ε, για παράδειγμα, θα έχετε ένα smartphone. Ένα τηλέφωνο Nokia, ένα τέτοιο smartphone για παράδειγμα που μπορώ να αγοράσω στις Βρυξέλλες, πολύ πιθανό να έχει ε, παρασκευαστεί, κατασκευαστεί στην Κίνα. Όμως είναι η μισή ιστορία. Πάνω από 50% της αξίας ε, του, ε, του προϊόντος δημιουργήθηκε στην Ευρώπη από σχεδιαστές και μηχανικούς η ικανότητα της Νόκια να διασφαλίσει αυτή την ε, αξία ε, εξαρτάται και από τα πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα σχεδιασμού. Αν τα, ε, τέτοιες, το έργο των επαγγελματιών μπορεί απλώς να αντιγραφεί, τότε έχουμε την απώλεια όλων αυτών των θέσεων εργασίας και στην Ευρώπη. Γνωρίζοντα αυτό, έχουμε δημιουργήσει ένα συνολικό, ολοκληρωμένο σύστημα για να προστατεύσουμε αυτά τα δικαιώματα και έχουμε και τα μέσα για να το κάνουμε. Επιλέξαμε να, να ε, προσπίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών στην ελεύθερη έκφραση και την προστασία δεδομένων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι ο υπέρτατος θεματοφύλακας ε, αυτών των ελευθεριών και ήδη αυτό επιβεβαιώθηκε μόλις αυτό το μήνα σε μία απόφαση ορόσημο ε, για την δραστηριότητα στο διαδίκτυο. Στόχος της ΑΚΤΑ είναι να επεκτείνει τα ωφέλη του συστήματος αυτού ε, και έξω από τα σύνορά μας. Είναι ένα μικρό αλλά και σημαντικό βήμα στη διαδικασία μας για την καταπολέμηση της πειρατείας και της παραποίησης. Ε, εκτιμούμε περίπου τον κύκλο εργασιών αυτής της ε, βιομηχανίας στα 200 δις ευρώ κάθε χρόνο. Και αυτό περιλαμβάνει οποιοδήποτε αντίγραφο ακόμα και αν το αντίγραφο πωλείται στη χώρα που ε, δημιουργήθηκε, κατασκευάστηκε, για παράδειγμα στην Κίνα. Δεν καλύπτει όμως τις πληροφορίες, δηλαδή τι είναι νόμιμο και τι παράνομο. Απλώς ε, ε, προσδιορίζει τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστούν οι παράνομες δραστηριότητε. Και ενθαρρύνει και την διεθνή συνεργασία μεταξύ 38 χωρών. Αξιότιμα μέλη, υπό τη δική σα ε, σύσταση, ένα από τα κύρια ε, επιτεύγματα τη Ευρωπαϊκή σε αυτή τη διαπραγμάτευση είναι ότι ε, βασίζεται στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματο η ΑΚΤΑ, δηλαδή του κανονισμού του 2004 για την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, τον κανονισμό τελωνική δράση κατά, την παραποίηση, κατά του 2003, οδηγία κοινωνίας ενημέρωσης του 2001 κλπ. Αυτές οι οδηγίες ε, καθορίζουν το δίκαιο ε, που προσδιορίζει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει για την προάσπιση τη ε, πνευματική ιδιοκτησία στην Ευρώπη. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν χρειάζεται να κάνει καμία αλλαγή στην υφιστάμενη νομοθεσία για να συμμορφωθεί με την άκτα. Ω εκ τούτου δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στην ε, ε, ισορροπία που υπάρχει μεταξύ δικαιωμάτων και δικλείδων ασφαλεία για του Ευρωπαίου πολίτε. Βεβαίω αυτό πρέπει να ε, το προσπίσουμε σε όλο τον κόσμο. Η άκτα επεκτείνει το επίπεδο ασφάλειά μα σε ένα ευρύτερο φάσμα και ελπίζουμε ότι αυτή η σφαίρα θα αποτελέσει θα επεκταθεί ακόμα περαιτέρω μετά την προσχώρηση και άλλων χωρών. Αυτά εν ολίγης ε, ως προς το περιεχόμενο της άκτα. Έχει υπάρξει δημόσιος διάλογος για αυτό το θέμα και γι' αυτό πρέπει να πω και τι δεν θα κάνει η άκτα. Παρά τα όσα έχετε ακούσει, η ίδια Η άκτα δεν θα λογοκρίνει το διαδίκτυο. Με αυτό ε, εννοώ ότι δεν θα ελέγχει τη δραστηριότητα των πολιτών. Δεν θα υποχρεώνει δεν θα επιβάλλει υποχρεωτικό έλεγχο των ε, ε, υπολογιστών ιδιωτών. Ας μην ξεχνούμε ότι το δίκαιο του ΠΟΕ προστατεύει και τα γενώσιμα φάρμακα, για παράδειγμα. Μετά από δημοκρατικές διαβουλεύσεις καταλήγουμε στα ίδια συμπεράσματα και νομίζω ότι στα ίδια κατα... συμπεράσματα θα καταλήξετε κι εσείς. Όλα αυτά εξηγούνται ξεκαθάρα και στο κείμενο της συμφωνίας. Υπάρχουν πολλές παρανοήσεις και σίγουρα θα τις συζητήσουμε εδώ σήμερα και σίγουρα ε, με περισσότερες λεπτομέρειες στο αυριανό εργαστήριο. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε ένα παράδειγμα που νομίζω ότι ε, είναι αντιπροσωπευτικό για τη σύγχυση που επικρατεί. Πολλά έχουν υποθεί σε ό,τι αφορά την ε, δημοσιοποίηση των δεδομένων των χρηστών. Αυτό έχει υποθεί ότι θα οδηγήσει στην παρακολούθηση ιδιωτών από ιδιωτικές εταιρείε. Αν δείτε όμω καλά την ε, συμφωνία, αλλάζουν τα πράγματα. Η Άκτα αναφέρει ότι οι χώρες που προσχωρούν δύνανται να δώσουν ε, στις ε, αρχές επιβολής του νόμου τη δυνατότητα να δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα εάν ο λογαριασμός αυτός ε, υπάρχει υποψία ότι, υπάρχει ότι χρησιμοποιείται για την παραποίηση, για παραβίαση της άκτα. Για να καταλάβετε ένα ενδεχόμενο σενάριο, για παράδειγμα, ε, ε, λέγεται ότι μια ιστοσελίδα δίνει πρόσβαση σε ε, παρανόμως ε, για να κάνει κάποιο download ένα επεισόδιο μια σειρά, για παράδειγμα. Τότε θα, θα μπορούσε το δικαστήριο, για παράδειγμα, μετά από απόφαση να ζητήσει ε, να, δημοσιοποιηθεί, να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία αυτού που εκμεταλλεύεται, που αποφελείται από την δραστηριότητα. αλλά γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει απόφαση και ε, να έχει, να έχει υπάρξει καταγγελία στι αστυνομικέ αρχέ. Όπω εγώ, για παράδειγμα, θα κατήγγειλα την ε, κλοπή ε, τη τσάντα μου, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει καμία διαδικασία χωρί ε, την απαραίτητη ε, νομική διαδικασία. Πρέπει να καταλάβετε όμως ότι δεν είναι εξίσου νομικά δεσμευτική. Λαμβάνει υπόψη άκτα και το εθνικό δίκαιο. Λέει λοιπόν ότι ενδεχομένω να ακολουθήσουν μια διαδικασία υπογράφοντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποχρεούνται να το κάνουν. Με αυτή τη διάταξη, η άκτα δεν αλλάζει τίποτα στην ελευθερία μα ε, για τη διαμόρφωση πολιτική. Απλώ ε, υποδεικνύει αυτό που ορισμένοι από, τις, ε, από, τα, από συμβαλόμενα μέρη θεωρούν βέλτιστη πρακτική. Για μα αυτό σημαίνει ότι εάν πάμε στα δικαστήρια για παράδειγμα για να για να ζητήσουμε την απαγόρευση της δημοσιοποίησης ε, ε, δεδομένων ε, ιδιωτών, αυτό μπορεί να γίνει και το κάναμε και σε οδηγία πριν από 15 χρόνια. Υπάρχει λοιπόν μια ισορροπία εδώ πέρα. Γιατί υπάρχει μια σειρά δικλείδων ασφαλείας για την προστασία των δικαιωμάτων των ιδιωτών και των χρηστών του διαδικτύου. Μόλις αυτό το μήνα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, εξέδωσε μια απόφαση ορόσημο. Το δικαστήριο είπε πολύ απλά ότι τέτοιοι πάροχοι υπηρεσιών όπως η Google ή το Facebook δεν δεν μπορούν να δημοσιοποιούν τα, τα δεδομένα των χρηστών και αυτή η απόφαση μας επιθυμίζει ότι μπορούμε να είμαστε ήσυχοι σε ό,τι φορά τα προσωπικά μας δεδομένα. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε κάτι το οποίο προβληματίζει πολλούς. Μπορούμε να πούμε ότι όλοι εδώ ξέρουν κάποιον που έχουν κατεβάσει το ε, ε, ε, ένα τραγούδι ή ένα επεισόδιο μιας τηλεοπτικής σειράς. Ε, δεν λέω ότι συμφωνείτε με αυτή την δραστηριότητα, αλλά για μένα δεν υπάρχει θήκη διαφορά από το να πάρουμε κάτι το οποίο δεν, δεν είναι δικό μας ε, πρακτικά και κάτι στον ψηφιακό κόσμο. Δηλαδή, δεν αποδίδουμε χρήματα που θα έπρεπε να αποδώσουμε στον δημιουργό. Ίσως κάποιοι στο πίσω μέρος του μυαλού σα ανησυχείτε ότι οι γνωστοί σας ενδεχομένω να ε, πάνε ακόμα και στη φυλακή ή τουλάχιστον να πληρώσουν πρόστιμα για αυτόν τον λόγο. Αλλά ο σημερινό νόμος είναι ξεκάθαρος εδώ. Γιατί είναι ποινικό αδίκημα που πρέπει να καταγγελθεί στην αστυνομία, αλλά ε, το να κατεβάζει κάποιο παρανόμος δεν είναι ποινικό αδίκημα. Ε, δεν υπάρχει λοιπόν ποινική δράση εκτός και αν αυτό έχει γίνει σε ε, εμπορική κλίμακα. Αν δηλαδή κάποιο ε, κερδοσκοπεί, κάποιο ε, όπω η Mega Upload και τώρα βρίσκονται στο, στο στόχαστρο του νόμου. Αυτό δεν αφορά του δεκάδε χιλιάδε ε, χρήστε ανά τον κόσμο. Αυτό είναι κοινή λογική και δεν αλλάζει με την άκτα. Αν αυτό είναι λοιπόν ένα από του λόγου που έχετε αμφιβολίε, Α είμαστε ξεκάθαροι. Δεν ποινικοποιούμε κάτι το οποίο δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα αυτή τη στιγμή. Ε, όλοι αυτοί οι νέοι δεν θα τους ε, στείλουμε στα δικαστήρια ε, για, για παραποίηση. Κάποιοι λένε ότι είναι αντιδημοκρατική η συμφωνία. Δεν αναθέτουμε εξουσίες σε κάποιον σκιώδη ε, μυστικό οργανισμό. Πρώτον συμμετέχουν όλα τα, τα κράτη-μέλη. Μετά, οποιασδήποτε τροπολογίε προτείνονται από την Επιτροπή, από τα κράτη-μέλη, πρέπει να περάσουν από πλήρη διαδικασία κύρωση υπό τι Ευρωπαϊκέ Συνθήκε. Δηλαδή, εσεί και τα Εθνικά Κοινοβούλια συμμετέχετε πλήρω στη διαδικασία. Η διαδικασία διαπραγματεύσεων υπήρξε επίση δημοκρατική. Το Κοινοβούλιο ήταν απολύτω ενήμερο ε, καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ε, Ιδίω από όταν ανέλαβα εγώ τα καθήκοντά μου, θεωρώ. Από τη στιγμή που ανέλαβα την υποχρέωση για αυτό το φάκελο, κάλεσα όλα τα διαπραγματευόμενα μέρη να ε, δημοσιοποιούν τα προσχέδια και αυτό και έγινε. Εσείς είχατε πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να παρακολουθείτε το έργο της Επιτροπής. Και λάβαμε υπόψη και όλα όσα μας έχει τυπήσει σε όλη τη διαδικασία. Τρία παράδειγμα σας δίνω. Πρώτον, η Επιτροπή δημοσιοποίησε όλο το κείμενο των διαπραγματεύσεων ε, το 2010. Δεύτερον, ακούσαμε τις ανησυχίες σας για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ε, ιδιωτική ζωή. Και ε, είμαστε σίγουροι πλέον ότι δεν υπάρχουν αλλαγές ε, στην ε, προστασία αυτού του τομέα. Αντιθέτως, συμπεριλαμβάνονται πολλές δικλείδε ασφαλεία και πολλά από αυτά τα ζητήματα υπόκεινται πλήρω στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ξεκινώντα από το κεφάλαιο των θεμελιώδων δικαιωμάτων και τρίτον, τα, τα γενώσιμα φάρμακα προστατεύονται πλήρω. Όμω, όλα αυτά αποκλείονται. Ε, ε, αποκλείονται από την άκτα όλα αυτά. Επιπλέον υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στην ε, δήλωση Ντόχα για τα γενώσιμα φάρμακα. Όλοι λοιπόν ε, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ευτυχείς με τα αποτελέσματα αξιότιμα μέλη. Χαίρομαι που υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ε, του κοινού για αυτή τη συμφωνία. Είναι ε, ε, ένδειξη υγεία η συμμετοχή των πολιτών. Όμω δυστυχώ δεν υπάρχει ακρίβεια σε αρκετού από αυτού του χειρισμού και είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό ότι αυτή η συμφωνία καταστρατηγεί τις βασικές αρχές, δημοκρατικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα περισσότερο με απογοητεύει ότι κάποιοι θέλουν ε, να υπερασπιστούν τις, ε, ε, τις ελευθερίες του διαδικτύου με το να επιτίθενται σε συγκεκριμένους ε, ιστοτόπους. Εγώ ήμουν δικηγόρος, ε, νομικά σπούδασα και εδώ και πάρα πολλά χρόνια προασπίζομαι τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Ε, συνέβαλα στην έκθεση Σπινέλη και κατέρτισα και το πρώτο εκατάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και συνέβαλα και εγώ με, το, με τη σειρά μου στη διαμόρφωση θεμελιώδων δικαιωμάτων στις συνθήκες Λισαβόνας. Και βεβαίως δεν θέλω να, ε, να διακινδυνευτούν αυτά τα δικαιώματα. Το Συμβούλιο αποφάσισε ομοφόνο να υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Κατανοώ βεβαίω ότι ε, για κάποιους δεν αντικούν τα όσα κάνω προσωπικά. Γι' αυτό συστήνω στους υπολείπους επιτρόπους να φέρουμε την άκτα ενώπιον του δικαστηρίου. Το δικαστήριο θα μας παράσχει την απαραίτητη ε, ασφάλεια δικαίου και η απόφαση θα στηρίξει και θα βοηθήσει για μια ήρεμη ε, και λογική συζήτηση που πρέπει να διαξάγουμε. γιατί πρέπει να σημειώσουμε πρώτος αυτό το θέμα. Κάποιοι μπορεί να πιστεύετε ότι τα οικονομικά ωφέλη δεν ε, αξίζουν τον κόπο. Όμως πρέπει να έχουμε μια καλή ε, στρατηγική διασφάλιση των δικαιωμάτων, των πνευματικών δικαιωμάτων, γιατί ζούμε σε μια εποχή ανταγωνισμού και δεν το κάνουμε εμεί, δεν το κάνει κανένα. Πρόεδρε, εξαιρετικά μέλη, σας καλώ να δείτε ε, με ευνοϊκή στάση αυτή την απόφαση. Ευχαριστώ. Thank you, You've got a Έχουμε πρόβλημα. σα ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Έχουμε πρόβλημα ότι φεύγουν οι διερμηνεί. Ή λοιπόν θα διακόψουμε εδώ τη συζήτηση και θα τη συνεχίσουμε αύριο ή θα συνεχίσουμε αγγλικά. Πράγμα που δεν μου φαίνεται δίκαιο να συνεχίσουμε συζητήσει σε μία και μοναδική γλώσσα. Παρακαλώ, λοιπόν, τον εισηγητή να μου πει ποια είναι η απόψη του. Δεν θέλω να κάνω παρατήρηση σε δύο λεφτά. Θέλω να έχω αρκετό χρόνο να παρουσιάσω την θέση του Κοινοβουλίου. Προτιμώ να το κάνουμε αυτά αύριο. Αύριο όμως στις 9 έχουμε συνέντευξη στο BBC. Και ε, εγώ και ο Επίτροπος δικού. Μπορεί να είμαστε όμως στις 9.30. Μετά να ψηφίσουμε τότε πρώτα και να το κάνουμε τη συζήτηση μετά την ψηφοφορία. Εσείς πρόεδρε αποφασίζετε μπορώ να ελευθερωθώ από τις 9.30 έως 12.30 το πρωί. Μπορώ να αναβάλω ό,τι ραντεβού είχα για αύριο το πρωί. Λοιπόν, μετά την ψηφοφορία, στις 10 θα αρχίσει η συζήτηση με αυτού του θέματος. Σας ευχαριστώ πολύ. It's good, <laughs>